Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν οι ομάδες ε, ξέρουν ότι έχουμε ψηφοφορία και ότι μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες και κάποιοι συνάδελφοι είναι απόντες. Αλλά αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες λοιπόν. Ε, τώρα οι απόντες ε, έχουν πάντα άδικο. Ο εισηγητής είναι εδώ για τους οργανισμούς. Θέλετε πως να πάρει το λόγο. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, γενική έκθεση για τους οργανισμούς. Όσον αφορά την εφαρμογή του προπολογισμού της Ένωσης ε, και τον οργανισμό της Ένωσης. Οπότε ξεκινάμε. Τροπολογία 1 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. λοιπόν, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη δύο, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Υπέρ παρακαλώ. Αντίρρηση. Συνολικά το κείμενο λοιπόν. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Λοιπόν, ε, περνάει. Τροπολογία. Η 4 έχει ε, ε υποσυρθεί. 5 υπέρ, κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 7 που είναι και, έχει και προφορική τροπολογία υπέρ, παρα, ε, κατά. Αποχέ. Α, είναι δύο τμήματα, με συγχωρείτε. Το πρώτο τμήμα, παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Αποχέ. Λοιπόν, να το ελέγξουμε γιατί δεν είδα τι γίνεται. Λοιπόν, εγκρίνεται, ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε, παρακαλώ, και το δεύτερο τμήμα, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει ο συσχετισμός. Ναι, απορρίπτεται. Η 7 έχει αποσυρθεί 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ α, α, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 συμβαστική 1 ε, α μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 έχει αποσυρθεί. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 δύο τμήματα ή μάλλον τρίτα, τρίτα τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 κατά πίπτη γιατί κρίθη 27, 28 λοιπόν υπέρ. Λοιπόν, να ελέγξουμε την 28 παρακαλώ.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 Λοιπόν, πέρασε Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 44 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλε 1 υπέρ κατά αποχές λοιπόν να την ελέγξουμε έμπλε 1 έμπλε 1 Πέρας, δεκτή. Έμπλε 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 4 ε, καλύπτεται. Έμπλ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπλ 6 καλύπτεται. Έμπλ 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 1 καλύπτεται. Λίμπε 2 δεν θα ψηφίσουμε. Λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπα 4 και 5 καλύπτονται 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 7 ε, συγγνώμη υπερκατά. Για να ελέγξουμε. Τη Λίμπε 6 λέει πρόεδρος. Α, όχι, τη Λίμπε 7 διορθώνει πρόεδρος. Ωραία. Πέρας. Δεκτή. Λίμπε 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συνολικά το ψήφισμα αποστροποποιήθηκε ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 18-3. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Οπότε τώρα. Ξεκινάμε τώρα τις επιμέρους προφορίες των οργανισμών. Με το 11 έισα την απόφαση για την απαλλαγή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε οι δύο καταπίπτει λοιπόν η απόφαση για την ε, απαλλαγή με ονομαστική η οποία έρχεται. Πέρας. 15 υπέρ 5 κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, για το ψήφισμα, γιατί σε αυτή την απόφαση συμπεριλαμβάνεται η, λοιπόν, το τροπολογία το ψήφισμα, τροπολογία 4, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, το ψήφισμα συνολικά ονομαστικά άρχεται. πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Ωραία, συγχαίρουμε τον συγκητή. Λοιπόν, Μπέρεκ. Απόφαση για την απαλλαγή. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά απόχέ. δεκτή. Οπότε καταπίπτει 2 η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απαλλαγή η οποία και άρχεται. Πέρας. 17-3. Ωραία. Ψήφισμα λοιπόν τώρα. 4 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 7 υπέρ, 7 και 8 υπέρ κατά αποχές, δεκτές 9 και 10 υπέρ κατά αποχές, δεκτές 11 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή και η 14 εντάξει ωραία 15 και 16 επίσης ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 17 και 18 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 19 και 20 υπέρ, ε, ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 21 υπέρ κατά αποχές α να ελέγξουμε ωραία ελέγχουμε την 21 Πέρας. Απορρίπτεται. 10-11. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περνάμε, περνάμε τώρα στην ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα η οποία και άρχεται. Πέρας. 19 ευχαριστώ πολύ. CDT. Τροπολογία 1 για την απαλλαγή πέρα κατά αποχέ εγκρίνεται. Η δύο ονομαστική τώρα για την απαλλαγή άρχεται. Πέρας 17-4. Ευχαριστώ πολύ. Ψήφισμα. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές. αποχε δεκτη 5 υπέρ κατά αποχέ. Δεκτή 6 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές λοιπόν να ελέγξουμε την 8 ελέγχουμε την 8 πέρας δεκτή η 9 που έχει και μια προφορική τροπολόγηση υπέρ κατά ε, απορρίπτεται ή θέλετε να το ελέγξουμε ε, ας ελέγξουμε. Την εννέα. Παρακαλώ ελέγχουμε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Α, μάλιστα. Α, οι σοσιαλιστές είναι κατά της προφορικής τροπολογίας, αλλά υπέρ του κειμένου. Λοιπόν, πρώτα ψηφίσουμε την ε, προφορική τροπολογία, παρακαλώ. Ψηφίσουμε πρώτα για την ορολική, ε, προφορική τροπολογία. Πέρας. Ωραία, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίσουμε το κείμενο συνολικά το ίδιο το κείμενο, χωρίς την προφορική τροπολόγηση. Με ηλεκτρονικό τρόπο. Πέρας. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 1 καλύπτεται κουλτ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 4 συμπεριλαμβάνεται 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή το ψήφισμα ονομαστική άρχεται περασε 19 19-3, ευχαριστώ πολύ. Σεντεφόπ. Στη Θεσσαλονίκη. 1 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. Οι δύο καταπίπτει. Ονομαστική για την απαλλαγή άρχεται Πέρας. 18-4. Ευχαριστώ πολύ. Το ψήφισμα λοιπόν τώρα. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 με την προφορική τροπολόγηση υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική υπάρχουν όπως και πριν η, η πλειοψηφία ήταν η ίδια οπότε την προϋποθέτω οπότε ψηφίζουμε το ίδιο το κείμενο του κειμένου είναι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές. τα 10 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Έμπλα 1 έως 5 περιλαμβάνονται. Έμπλε 6 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 7 και 8 καλύπτονται. Ονομαστική τώρα για το ψήφισμα. Άρχεται. Λοιπόν, ε, ένα δεν ψήφισε. Λοιπόν, πέρασε. 18 18-3 ευχαριστώ πολύ. Σέπολ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. Οι δύο καταπίπτει. Η απόφαση για την απαλλαγή ονομαστική άρχεται. Πέρας. 17-5. Ψήφισμα. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Συγγνώμη. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται 11 υπέρ. Κατά απο... Α... Λοιπόν, να ελέγξουμε την 11. Ελέγχουμε την 11. περα Απορρίπτεται 8, 15, 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 13. Υπάρχει προφορική τροπολόγηση, υπάρχει αντίρρηση. Ωραία, το κείμενο όσο έχει υπέρ, κατά Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. Την 14 παρακαλώ. Πέρας. Δεκτή. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Λίμπε 1 έως 4 συμπεριλαμβάνονται. 5 υπέρ. Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχέ δεκτή. Λίμπε 6 υπέρ κατά αποχέ δεκτή. 7 έω 9 καλύπτονται 10 υπέρ. Λίμπε 10 υπέρ κατά αποχέ δεκτή. Το ψήφισμα συνολικά ονομαστική άρχεται. Πέρας. 21 προς 3, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ΕΑΣΑ. Ένα, υπέρ. Κατά δεκτή. Η δύο, ήταν ε, ταυτόσιμη τρία. κατά πίπτη. Ψηφίζουμε την απαλλαγή ονομαστικά άρχεται. Πέρας. 24. Ωραία. Ψήφισμα. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά αποχές. Λοιπόν, μάλλον περάσαμε αλλά να την ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 9. Α, υπαρχει άλλο ένα, ένας. Ωραία, εγκρίνεται. 12-11. Λοιπόν, 10, προφορική τροπολόγηση, υπάρχει αντίρρηση, ωραία, το κείμενο ω έχει υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Να το ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε. Την 10. Εγώ νομίζω πως θα είναι ο ίδιο σχετισμός με πριν, αλλά τέλος πάντων, να σε ελέγξουμε. Α, ένας δεν ψήφισε. Ωραία. Δεκτό. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές. Λοιπόν, να την ελέγξουμε. 12. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές. Λοιπόν, να την ελέγξουμε. Να την ελέγξουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι σαφή τα πράγματα. Πέρας. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τραν 1 έως 3 καλύπτονται. Τραν 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τραν 5-6 καλύπτονται 7, τραν 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τραν 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τραν 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τραν 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τραν 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τραν 12 και 13 καλύπτονται, ονομαστική, τελική για το ψήφισμα, άρχεται. Πέρασε. Λοιπόν, 21-3 εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Εάσο. Λοιπόν, εδώ δεν υποβλήθηκε καμία τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε απευθείας ονομαστικά για την απαλλαγή. Όποιος είναι υπέρ της απαλλαγής θα ψηφίσει υπέρ. Και όποιος είναι κατά, κατά, ονομαστική. Πάμε, άρχεται. Πέρας λοιπόν. 21-3. Ευχαριστώ πολύ. Ψήφισμα. 1 υπέρ. Κατά αποχέ δεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχέ. Λοιπόν, ελέγχουμε τη 2. Ελέγχουμε τη 2. Πέρας. Δεκτή. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και την 3. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πέρας. Δεκτή. Εδώ είμαι σύμμογο να μετάσχει προσφυγή. 4. Υπέρ. Κατά Δεκτή. 5. Υπέρ. Κατά Δεκτή. 6. Υπέρ. Κατά Δεκτή. 7. Υπέρ. Κατά Δεκτή. 8. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λίμπε 1 και 2 καλύπτονται. Λίμπε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λίμπε 4 καλύπτεται. Λίμπε 5. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Λίμπε 6 Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Λίμπε 7 και 8 καλύπτεται. Και συνολικά το ψήφισμα. Ονομαστική άρχεται. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με την ΕΑΣΟ. E Η ECR μου το τόνισε. Το ECR. Στο κατάλογο ψηφοφοριών λέγεται το συν είναι να αναβληθεί και το μείον είναι να χορηγηθεί. Θα πρέπει να επαναλάβω την ψηφοφορία. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείτε ε, ε, ανάποδα. Όποιο θέλει απαλλαγή, να δοθεί απαλλαγή, πρέπει να ψηφίσει κατά οποίο δεν θέλει να δοθεί, συγγνώμη, συγγνώμη είπα το, το αντίθετο. Λοιπόν, να ξαναψηφίσουμε για την απαλλαγή παρακαλώ. Η κυρία Γιάννα μιλάει στεχώς χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία που κάναμε. Γιατί δεν υπήρχε το υποβληθή τροπολογία. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν πρόσεξα. Λοιπόν, αν θέλετε να αναβληθεί η ψηφοφορία, τότε πρέπει να ψηφίσετε υπέρ. Συν. Συν. Εντάξει. Αλλά το ECR ακριβώς, εγώ είπα το αντίθετο από ό,τι γράφει εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία γιατί έκανα λάθος. Το παραδέχομαι. Εγώ φταίω. Λοιπόν, συν σημαίνει αναβάλλεται και μείον σημαίνει χορηγείται. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την απόφαση για την απαλλαγή. Εντάξει. Συνεχίζει η κυρία Γιάλα χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, ε, με συγχωρείτε το ανήγγυλα διαφορετικά. Το ανήγγυλα διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Θα πρέπει να ξανακάνουν την ψηφοφορία γιατί την ε, παρουσίασα λάθος. Αν ψηφίζετε συν, πράσινο, θέλετε να αναβληθεί η απαλλαγή. Εντάξει, αυτό ψηφίζουμε τώρα. Το ECR μου το τόνισε ότι δεν κατάλαβαν. Όπως σου παρουσίασα υπήρξε παρανόηση. Με συγχωρείτε. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν όποιο θέλει να αναβληθεί θα ψηφίσει συν. Όποιο ψηφίσει μείον δεν θέλει να αναβληθεί. Η χορήγηση απαλλαγή. Λοιπόν, παρακαλώ ψηφίστε. Δεν ψηφίσατε ακόμη όλοι αυτό. Λοιπόν, ε, πέρας. Λοιπόν, ομόφωνα. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και με συγχωρείτε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Έμπα. Αρχή ε, ψηφίστηκε, ψηφίστηκαν όλα και το ίδιο το ψήφισμα. Έγινε, ολοκληρώθηκε η τελική ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε η τελική ψηφοφορία, έτσι δεν είναι. 20 προς 4. προς 4. Εδώ, εδώ. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ένα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση για την απαλλαγή. Άρχεται η ψηφοφορία. Εδώ είναι ανάποδα. Όσον αφορά την απλούστευση και εγώ θα είχα ορισμένε ε, προτάσεις. Πέρας. 24. Ευχαριστώ πολύ. Χορηγείται η απαλλαγή. Και θα έρθουμε στο απολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 7 υπέρ, καταπίπτει 8 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση για την 8. Πέρας. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 10. Πέρας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 ε, η προφορική τροπολογία και συνέχεια το ίδιο το κείμενο υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 1 καλύπτεται έκον 2 έως 5 ε, και 6 on block. 2 μέχρι 6 πέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 7 καλύπτεται 8. Πρώτο τμήμα καλύπτεται το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. ένας. 20 προς 4 εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην ε, πρόληψη ε, των νόσων υπερ... Ένα. Οι δύο... Ε, η, η απόφαση για την ε, απαλλαγή άρχεται. Πέρας. 21 προς 3. Ευχαριστώ πολύ. Στο ψήφισμα 4. Πέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 πέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 πέρ κατα κατά αποχές εγκρίνεται MV1 καλύπτεται MV2 έως 4 μπλοκ 1 έως 8 MV μπλοκ. δεν υπάρχει αντίρρηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 9 έως 12 καλύπτονται τελική ψηφοφορία ονομαστικά τη ψηφοφορία Πέρας. 21 προς 3. Η Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 19-5, ευχαριστώ. Το ψήφισμα. 3 υπέρ κατά, αποχές, να το ελέγξουμε, θεωρώ ότι εγκρίνεται, αλλά έλεγχος. Η τρία, έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 13-10 δεκτή.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 1 έως 4, ωραία. 1 έως 4 unblock. μέχρι 3, 1 έως 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 έως 12 υπέρ. Unblock, υπέρ. Όχι. 4-5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 ναι επέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 επέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 επέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 προς 4. Ευχαριστώ πολύ τώρα. Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Περιβάλλοντος στην Κοπενχάγη. 21. Ε, σημείο 21. Τροπολογία υπερθυμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση να χορηγηθεί από αλλαγή ονομαστική άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα το ψήφισμα 4 υπέρ κατά υπέρ της 4 Ε, ψηφορία διεξάγεται όταν όλοι κάνουμε το ίδιο ταυτόχρονα. Λοιπόν, ας ελέγξουμε την 4. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να καταλάβω, να δω. Ωραία, λοιπόν, απορρίπτεται. Ευχαριστώ. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, θα, τα, θα ελέγξουμε την 5. Ωραία. Πέρασε του ελέγχου της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εγώ ήθελα να πω ότι ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, τελικά δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. 6 κατά πίπτη. 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 9, ε, προφορική τροπολογία, υπάρχει αντίρρηση, το κείμενο υπέρ κατά εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 ΕΠΕΡ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 ΕΠΕΡ, κατά αποχές εγκρίνεται 13 ΕΠΕΡ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η μία και οι δύο καλύπτονται. Μπορούμε δεκατρία μπορούμε να το ελέγξουμε. Κατά την άποψή μου απορρίπτεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Το σύστημα είναι πολύ βραδύ. Λοιπόν, εγκρίνεται, λυπάμαι λέει πρόεδρος, ωραία. Έμβη 1 και 2 ε, καλύφθηκαν, Εκαλύφθηκαν 3 και 4 μπορούμε αν μπλοκ υπέρ κατάποχες εγκρίνεται 5, έμβη 5, το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 και 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τώρα το ψήφισμα συνολικά ονομαστικά έρχεται Προς προς 3 ευχαριστούμε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου τη Αλία, σημείο 22, τροπολογία υπερφών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση θα χορηγηθεί από αλλαγή ονομαστικά έρχεται. Πέρας. 24 ευχαριστώ. Το ψήφισμα. 4 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 5 υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση έλεγχος για την 5. Η 5. εγκρίνεται 6 περιφερειακή ευρωπολογία, υπάρχουν αντιδρήσεις και το κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε unblock πες 1 έως 6 έως 14 Ω 10 εντάξει 1 έως 6 πες 1 έω 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 έως 12, 9, 9 συγγνώμη, 9 και 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 ε, υπέρ, κατά αποχές, ε, έλεγχος για την 11. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. 11, πες 11 απορρίφθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση έλεγχος γιατί 14 πιστεύω ότι έγινε δεκτή 14 πέρας εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστικά Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 21-3. Ευχαριστώ. Εύσα. Ε, Ευρωπαϊκή. Ένα υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ψήφος για τη χωρίς απαλλαγής ονομαστικά άρχεται. Πέρας. 19-5. Ευχαριστώ. Το ψήφισμα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 Έλεγχος για την 21. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. 22 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έγινε δεκτή. Έλεγχος για την 23. εγκρίνεται σαφώς 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 30 να γίνει έλεγχος για την 31 για να είμαστε σίγουροι πέρας απορρίπτεται λυπούμε λέει πρόεδρος 32 υπέρ Α, ωραία, να γίνει έλεγχος για την 30 επίσης, 30. απορρίπτεται ισοψηφία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται MV1 έχει καλυφθεί μπορούμε να ψηφίσουμε κάποιες unblock όλες οι 2 ως την 11 unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ονομαστικά το ψήφισμα στο σύνολό του 24. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το... Ε, η απόφαση για την απαλλαγή ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. 19.5. Ευχαριστώ. Το ψήφισμα 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 4. πέρας απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ όχι 6 υπέρ Οχτώ υπέρ, οχτώ Ψηφίσαμε την 6. Ναι, εγκρίθηκε. Ωραία. Η 7 καταπίπτει 8 λοιπόν. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση, έλεγχο για την 9. Νομίζω ότι καταψηφίστηκε, αλλά ας το ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 με προφορική τροπολογία που απορρίφθηκε το ίδιο το κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ A, ε, B μέχρι το 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Το ψήφισμα ονομαστικά. Πέρας. 24 ευχαριστώ. ΑΙΟΠΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση χωρίς απαλλαγή, ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. προς ευχαριστώ. Το ψήφισμα 4 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος για την 4 παρακαλώ. Εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 8 υπέρ. Παρακαλώ. Ωραία, να γίνει έλεγχος για την 5. Εγώ βλέπω όσους ψηφίσουν από πίσω από σένα. Κρίθηκε. Λυπούμε. Οχτώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εννέα με προφορική τροπολογία που δεν έγινε δεκτή, το κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 11. Πέρας εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον το πρώτο τμήμα έχει καλυφθεί το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπορούμε να γίνουμε όλες ε, να γίνουν μπλοκ όλες οι τροπολογίες έκον 2 σε 6 2 ως 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται έκον 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα το ψήφισμα ονομαστικά έρχεται. Πέρας. 20 προς 4, ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας Τεχνολογίας 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η απόφαση χωρίς απαλλαγή ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία.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 Απορρίπτεται. Τώρα το ψήφισμα ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 προς 3. Ευχαριστώ. ΕΜΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απόφαση χρήσης απαλλαγής ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. 19 προς 5 το ψήφισμα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές θα μπορούσε να απορριφθεί έλεγχος για την 7 παρακαλώ 7 Πέρασε. Απορρίπτεται 8 υπέρ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 εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 21 Πέρας. Α, όχι, το σύστημα είναι αργό. Ωραία. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές. Κατά την άποψή μου έγινε δεκτή, αλλά να γίνει έλεγχος για την 22 παρακαλώ. εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV4 μπορούμε να κάνουμε unblock τις τροπολογίες της MV όχι MV 4 μπορουμε να κανουμε unblock τις τροπολογιες της mv οχι mv 4 ως 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. 19-4. Τώρα, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών. 1. Υπέρ κατά Η αποφάση χωρί απολαγής ε, ονομαστικά άρχεται. Πέρας. 20 προς 4. Το ίδιο το ψήφισμα Τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ. Α, με, ε, υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία του ίδιου το κείμενο υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Το κείμενο ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. περασε Ένα υπέρ. Απόφαση χορήγησης απαλλαγής. Είκοσι Πρώτη συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 κατά πίπτη, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 10 προφορική τροπολογία. 11 ε, εγκρίνεται η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 4 υπέρ τα αποχέ εγκρίνεται. Τραν 6 έω 6, 7, 8 εγκρίνεται. Το κείμενο τώρα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφορία. The vote is closed. 20... Πέρασε. 24. Ενίσα 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφορία για την απαλλαγή Closed, 24. Ψήφισμα 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6. Ναι, ναι, ναι, 5, 5. Δεκαεπτά, δεκαεπτά. Έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για το 7. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά έλεγχος για το 16 νομίζω απορρίπτεται αλλά να δούμε απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 17 εγκρίνεται με σαφή διαφορά το σύνολο του κειμένου ονομαστική mm. 21 to 3. Thank you. The Railway Agency, Amendment 1, in favor. Οργανισμό Σειροδρόμων 1. Υπέρ καταβολή δεν εγκρίνεται. Και τώρα απαλλαγή με γνωστή ψηφορία ψηφίζουμε. The vote is closed, 20 to 4. And we have the... 24 εγκρίνεται. Το ψήφισμα αυτό εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε ηλεκτρονικό έργο για το 8 νομίζω εγκρίνεται. Εγκρίνεται ναι με μία ψήφο διαφορά. 9 υπέρ κατά άποχέ εγκρίνεται. 10 προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά. 11 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για το 14. 14. Check Και εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Έλεγχος και για το 15. Εγκρίνεται. Όντω. Τραν 2. κάνουμε όλε μαζί. 2 με 15. Τραν 2 με τραν 15. Δεν είχατε καμία αντίρρηση αποχέ. εγκρίνονται. Και τώρα το σύνολο του το ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Λείπει μία ψήφος. Πέρας. 23. Ευχαριστώ. Αρχή αξιογράφων και αγώνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση της απαλλαγή με ονομαστική ψηφόρια. 19.4. Τροπολογία 4 του Σεύρνους υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Για το 5 τώρα. <clears throat> Για το 5 έλεγχο. Στο ψήφισμα είμαστε. Τροπολογία 5. Πέρασε. Εγκρίνεται και τώρα 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά Έλεγχος επί του 9. Και απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Με προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για το 13 και εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ όχι 14 14 έλεγχος του 14 Πέρας. Ε, και εγκρίνεται. 15. Υπέρ κατά αποχές. 16. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Έλεγχος για το 16. Πέρας. Και απορρίπτεται. 17. Υπέρ. 8. Ε, συγγνώμη, υπερκατά? η ίδια πλειοψηφία και μπορείτε 18. 18 υπερκατά κατά εγκρίνεται. Έκον 1 με, όχι, έκον 2 με 4 υπερκατά αποχέ εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος πάλι. περασε 184. Σας ευχαριστώ και τώρα το ETF Ίδρυμα Εκπαίδευσης Επαγγελματικής Περκατά εγκρίνεται η απόφαση της απαλλαγής ονομαστική ψηφορία ψηφίζουν. Το 33, το, ε, το 33 της Μέσης Διατάξεως, ETF, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εκπαίδευσης. 19-4 το ψήφισμα τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 4 και εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά, έλεγχος. Και απορρίπτωση. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για το οκτώ. Απορρίπτωση. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10. Με την προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος 12. Έγκρινεται. Έμπλ. Όλες μαζί. Δύο με επτά. Όχι. Όλες μαζί. Δύο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα εγκρίνεται. Καλύπτεται το σύνολο τώρα του κειμένου και του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε πέρας ψηφορίας εγκρίνεται 21-3 EU Λίζε το 34 δηλαδή υπέρ κατά αποχές για το πρώτο τροπολογία εγκρίνεται η απόφαση απαλλαγής η νομαστική ψηφοφορία πέρασε 19, 4. Το κείμενο του ψηφίσματο τροπολογία 6. Υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 12 νομίζω ότι εγκρίνεται εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ αποχές εγκρίνεται 18 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 19 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 20 υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε όλες τις λίμπε 4 με 13 υπερκατά αποχές εγκρίνονται όλο το κείμενο με ονομαστική Πέρας 22. Το, 10, το 35. Όσα. οργανισμό ασφάλεια και Συνεργασία. Ε, η, η, απόφαση της απαλλαγής με νομιστική ψηφοφορία. Πέρας. Το ψήφισμα. Ψήφισμα το 4. Υπέρ κατά άποχες. Έλεγχος του 4. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για το 5. Έλεγχος για το 5. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για το 8. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το 9 απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά έλεγχος για το 12. Απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές έλεγχος και για το 13. Απορρίπτεται. Μεγάλη πλειοψηφία. 14 χωρίς προφορική τροπολογία, το κείμενο, εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Να κάνουμε όλες τις τροπολογίες έμπλ μαζί. Συμφωνείτε, ναι. Όλες μαζί. Υπέρ κατά αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα το συνολό του κείμενου του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 21. 3 οργανισμό εφοδιασμού τη Ευρατόμ ε, το 36 δηλαδή και εγκρίνεται η προτροπολογία και τώρα η απαλλαγή ονομαστική Πέρας. 24 ευχαριστώ δεν έχουμε κάποιο ε, κάποια διάταξη τροποποίηση, αλλά το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία Πέρασε. 21-3. Eurofund, δίδραμε για τη βελτίωση των διαβίωση και εργασία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται η πρώτη απολογία. Τώρα η απόφαση απαλλαγή με ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρα. Η 21. 3 εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του ψηφίσματο. Υπέρ. Κατά. Mm. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά α, αποχές έλεγχος για το 6. Α, απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά έλεγχος για το 11 ε, και εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες τις τροπολογίες έμπλε μαζί, μάλιστα. 2 με 7 δηλαδή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου του ψηφίσματος ονομαστική ψηφορία. Πέρασε. Ή 21-3. Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, Eurojust. Τροπολογία υπέρ κατά. Εγκρίνεται ονομαστική ψηφορία για την απαλλαγή υπέρ. Ε, κατά τέλος ε, ψηφίζουμε 24. Εγκρίνεται το ψήφισμα τώρα. 4 υπέρ κατά αποχές. Είναι το 5 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται έλεγχος για το 5. 5 έλεγχος. Ναι, έγκρινεται με σαφή πλειοψηφία. 6 υπέρ κατά Έγκρινεται 7 υπέρ κατά Έγκρινεται 8 υπέρ κατά αποχές. απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 10. Καταπίπτει. 11 υπέρ κατά Εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 13 υπέρ κατά Α, αποχές, έλεγχος. 13. Εγκρίνεται. 14 έχω την προφορική τροπολογία, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά. Έλεγχος για το 18. υπέρ Και εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες τις λίμπε μαζί 4 μέχρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται το ψήφισμα ονομαστική. Πέρασε. 29-3. 21-3 εγκρίνεται. 39 όλα 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το ψήφισμα, η απόφαση για την απαλλαγή ονομαστική άρχεται. Πέρασε. 24. Το ψήφισμα. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή 6 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή 7 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 8. Απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά οχές να ελέγξουμε την εννέα δεκτή 10 υπέρ κατά εποχέ. δεκτή 11 υπέρ κατά την ελέγχουμε δεκτή συγγνώμη 12 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε συγγνώμη συγγνώμη αλλά δεν δείχνουν όλες οι ομάδες ε, ποια είναι η πρόθεση τους απορρίπτεται σαφώς απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε και την 16. Σαφώς δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 18 χωρίς προφορική τροπολόγηση. Υπέρ του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές. Δεκτό. 19 υπέρ κατά αποχές. Δεκτό. 20 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 21 υπέρ. Υπέρ έλεγα κατά αποχές. Λοιπόν, να την ελέγξουμε παρακαλώ. Σαφώς δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 1 έως 5 μαζί. Λίμπε 1 έως 5 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Λοιπόν, και το ψήφισμα ε, ονομαστική άρχεται. Πέρας, 21-3. Ευχαριστώ πολύ. Ε, οργανισμό για θεμελιώδη δικαιώματο προηγεί είναι υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. Η απόφαση χορήγηση απαλλαγής σε ονομαστική άρχεται. Πέρας, 21 προς 3. Το ψήφισμα τώρα. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, λίμπε 5 και 7 μαζί μπορούμε. Υπέρ κατά αποχές δεκτές το κείμενο με ονομαστική άρχεται. Πέρας. 21-3. Εγκρίνεται. Frontex. Σημείο 41. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτό. Επόφαση απαλλαγής. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. 19 προ 4. Το ψήφισμα τροπολογία 5. Υπέρ κατά απόχέ, δεκτό. 6 υπέρ κατά απόχέ, δεκτό. 7 υπέρ κατά αποχέ. 7 έλεγα. Δεκτό. 8 υπέρ κατά αποχέ. δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχέ δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχέ, δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχέ. Α, να ελέγξουμε. Την 11. Την 11. Δεκτή. Οι δύο της Λίμπε, 4 και 7, 4 έως 7. Ωραία, υπέρ. Κατά αποχές, δεκτές. Το ψήφισμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. 20 προς 2. GNSS. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Η απόφαση απαλλαγής. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. 19 προς 5. Το ψήφισμα. 4 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8. 7 λέει η πρόεδρος. 7 δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε την 9. Ναι, να την ελέγξουμε παρόλα αυτά. Σαφώς ακρίθηκε. Δεν ήταν και τόσο σαφώ, ε, αλλά παρόλα αυτά εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ονομαστική για το ψήφισμα άρχεται. Πέρασε. 20 προς 4 ψήφοι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ψηφίσαμε για τους οργανισμούς και παρακαλώ να είμαστε πειθαρχημένοι για να προχωρήσουμε. Κανένα δεν αρέσουν βέβαια όλα αυτά. Λοιπόν, 51 58. Ο εισηγητής είναι ο Μάρκο Βάλλη. Θέλει να πάρει το λόγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, πρέπει να ψηφίσουμε για τα κοινά εγχειρήματα. Πρέπει να ψηφίσουμε για τα κοινά εγχειρήματα. Ναι, joint undertakings. 43 έως 50, 50 συγγνώμη, τα σημεία της 43 έως 50 έχετε όλα τα χαρτιά. Καταλαβαίνετε τι ψηφίζουμε. Ο συγκητής είναι ο Brian Hayes. Θέλει το λόγο. Όχι. Ωραία. Ωραία. BBI. Η βιομηχανία που βασίζεται στην βιολογία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η απόφαση χορήγηση απαλλαγή ονομαστική άρχεται. Πέρας. 20 προς 3. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το ψήφισμα. 2 υπέρ κατά αποχές. Δεκτό. 3 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 4. Πέρας. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. 20 προς 2. Λοιπόν, καθαρό ή αέρας, ε, καθαρός αέρας, ε, ε, η ουρανή δηλαδή, η ε, τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, ονομαστική για τη χορήγηση απαλλαγή. Πέρα, 20 προς 4. Και τώρα το ψήφισμα. 2. Οι 2 και 3. Δεν χρειάζονται να ψηφιστούν. Οι 4 υπέρ κατά αποχέ, δεκτή. Οι 5 υπέρ κατά αποχές, δεκτή το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. 20 προς 3. Δεκτή. Δεκτό το ψήφισμα. Excel ε, κοινό εγχείρημα τροπολογία ή ένα και δύο ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Η απόφαση απαλλαγής ονομαστική άρχεται. Πέρας. 18 προς 6. Το ψήφισμα. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Οπότε το 8 καταπίπτει 9. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. 10. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. 20 προς 4. Λοιπόν, τα στοιχεία καυσίμων και το υδρογόνο 2, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Η απόφαση απαλλαγής, ονομαστική, άρχεται. Πέρας. Δεκτό, δεκτή απαλλαγή 19-4, το ψήφισμα 2 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή 3 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή 4 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή 5 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή 6 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή 7 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή 8 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Περνάει 21-3. Ήμι. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η απόφαση απαλλαγή ονομαστική άρχεται. Πέρας. 20 προς 4. Ψήφισμα. 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 5. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή το ψήφισμα ονομαστική άρχεται πέρας 21-3 ευχαριστώ Λοιπόν, σύνδεξη για ενέργεια, ίτερ, ε, τροπολογία 1, η 1, 2 και 3, ε, ταυτόσιμες υπέρ κατά απορρίπτονται. Η απόφαση χορήγησης απαλλαγής, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Χορηγείται 23, ευχαριστώ πολύ, το ψήφισμα. Λοιπόν, α όχι, όχι, 6 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται, 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 8 πέρας απορρίπτεται 9 υπέρ κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 11 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Ίδια ισοψηφία. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 11 λέει η πρόεδρος. Α, με συγχωρείτε, τη 12, ναι, τη 12, ναι. Ελέγχουμε τη 12. Τη 12. Τη 12. Είναι τόσο χρωματιστή η εικόνα, αλλά απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. 13 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. 18-6. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Η απόφαση απαλλαγή ονομαστική άρχεται. Πέρα. Χορηγείται 20 προς 4. Το ψήφισμα. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχέ. Δεκτό. 3. Υπέρ. Κατά αποχέ. Δεκτή. Λοιπόν, τις τραν μπορούμε να τις κάνουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Όλες μαζί. Μέχρι τη 15. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κατά αποχές δεκτές. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. 21-3. Shift to rail. Το 50 δηλαδή. Το σημείο 50. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η απόφαση απαλλαγής ονομαστική άρχεται. Πέρας. 18-6, ευχαριστώ πολύ. Το ψήφισμα. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή 3 υπέρ. Κατά αποχές. Α, όχι, να ελέγξουμε την 3. Νομίζω ότι εγκριθήκε, αλλά... Εγκρίθηκε. 4 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά... Να ελέγξουμε την 5. Δεκτή σαφώ. 6 υπέρ. Κατά αποχέ. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά αποχέ. Δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχέ. Δεκτή. Λοιπόν, τι ε, τροπολογίε τραν όλε μαζί, εντάξει. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία. Όλε τι τραν. 6 με 14 υπέρ, κατά αποχέ, δεκτέ. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Δεκτό 21-3. Λοιπόν, για του άλλου οργανισμού 51-58 σημεία τη ημερήσια διάταξη συγητή ο κύριο Βάλλη. Και θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω του ε, συγητέ, λέει ο Βάλλη, για τη δουλειά. Δουλέψαμε καλά και καταλήξαμε σε εύστοχου συμβασμού. Υπάρχει ένα πρόβλημα για κάποια τροπολογία. Για μένα αυτό είναι κόκκινη γραμμή, είναι κάτι που αφορά την Άλντε ε, όσον αφορά κάποιο είδους ενιαίο κείμενο απαλλαγής ε, και έχει σχέση με την αποχώρηση της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και αυτό. Να δούμε τι θα ψηφίσουμε και εγώ θα αποσύρω την υπογραφή μου από το σχετικό κείμενο γιατί διαφωνώ. Ναι. Α, Μαρτίνα. Εγώ είμαι κατά της τροπολογίας. Θέλουμε την προφορική τροπολογία, λέει Μαρτίνα. Όχι, όχι, όχι, δεν, δεν κατέβασα τροπολογία. Είναι προσωπική μου άποψη. Κύριε Σαλαφράγκα, όχι μην το συζητήσουμε όμως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς να σας πω ότι έδειξε πολύ καλή διάθεση ο εισηγητής για να καλύψει όλα όσα θέλαμε οι πολιτικές ομάδες. Όταν υπάρχει καλή πίστη τα βρίσκουμε. Κρίμα θα ήταν μετά από όλη αυτή τη δουλειά του να μην προσυπογράψει την ε, έκθεση. Αυτή είναι η απόψή μας. Μα γιατί να μην κάνουν όλοι μια προσπαθιούλα και έτσι όλοι τελικά να είμαστε ικανοποιημένοι με την ε, έγκριση της έκθεσης. Τώρα είμαστε στην ψηφοφορία. Δεν θα ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση για το κείμενο τη διαπραγματεύσει. Αυτά πρέπει να έχουν γίνει προηγουμένω. Εντάξει. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε και θα δούμε πώς, ε, τι θα προκύψει τελικά. Ξεκινάμε με την ε, υπηρεσία εξωτερική δράση, το σημείο 51 τη ημερή διάταξη, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά απόχέ απορρίπτεται. Τρία υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. Περνάμε στην απόφαση. Για την απαλλαγή λοιπόν. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. 19 προς 3. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 7, υπέρ. Κατά. Λοιπόν, να την ελέγξουμε. Την 7, παρακαλώ. Ελέγχουμε την 7. 7. Πέρας, απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 10. 10. Πέρας, απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχέ, δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά ελέγχουμε την 15 Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. Mm μετά έχουμε την προφορική τροπολόγηση. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από ό,τι βλέπω στην προφορική τροπολόγηση. Άρα για το κείμενο μαζί με την προφορική τροπολόγηση. Υπέρ, κατά, αποχές. Ακριβώς λέει Λοιπόν, είναι το κείμενο μαζί με την προφορική τροπολογία. τι ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι, όχι, όχι, έλεγχος. Λοιπόν, δεν έχουν ψηφίσει όλοι ακόμη. Ε, είναι τόσο αργό το μηχάνημα. Δεκτή. 21 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Α, η 34 με την προφορική τροπολόγηση της. Υπάρχουν αντιρρήσει. Α, έχετε αντίρρηση. Οπότε το αρχικό κείμενο της 34. Χωρίς προφορική τροπολόγηση υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. 34 το αρχικό κείμενο χωρίς προφορική τροπολόγηση. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Το μηχάνημα μετράει ακόμη. Πέρας. Δεκτή, 12, 9. Απορρίπτεται λοιπόν πρόεδρος. Υπέρ, κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, το διορθώνει πρόεδρος. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε και αυτήν. Την 35. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά απόχέ, δεκτή. 44 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, πρώτο τμήμα τη 46. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο τμήμα. Όχι, 46, 46, συγγνώμη, 46, δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 46. Το δεύτερο της 46. Πέρας απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε. Άφετ 1. Όχι, άφετ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αφετ 3, αφετ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφετ 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφετ 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφετ 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρασε. Ε, συγγνώμη, άρχεται. Πέρασε. 20 προς 3, ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στο σημείο 52 της της διάταξης. Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τροπολογία 1 έως 4 που είναι ταυτόσιμες. Θέλουν να αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές θεκτές. Περνάμε στην απαλλαγή ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. 22 προς 1. Ε, Οπότε προτείνει η Κοντ να αναβληθεί η χωρίς απαλλαγή. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο ψήφισμα. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτό, δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές 8 υπέρ κατά αποχές δεκτό 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στην 11 χωρίς προφορική τροπολογία το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 12. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Ε, καταπίπτει βέβαια, καταπίπτει βέβαια το δεύτερο τμήμα άμα απορριφθεί το πρώτο. 13 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά ας ελέγξουμε. Α, είναι το θέμα του Brexit. Α, μάλιστα. Μάλιστα. 15 προς 6 λέει η πρόεδρος, συγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές, δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. Το ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. 21 προς 1 ψήφι και μία αποχή. Ε, με συνέδριο. Τροπολογίες 1 έως 3 και 4 για να δοθεί απαλλαγή. Ε, υπέρ εγκρίνονται. Οπότε η 3 καταπίπτει. Ψηφίζουμε όμως τώρα τελικώς ηλεκτρονικά. Άρχεται.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 νομίζω ότι έχει ενδεκτό, αλλά πέρας του ελέγχου εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ, καταπίπτει 14 με ψηφοφορία κατά τα πρώτα τμήμα απορρίπτεται και 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Α υπέρ κατά εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 18. 18 έλεγχος. Απορρίπτεται. 19. Με προφορική τροπολογία υπάρχουν ενστάσεις, άρα μόνο το κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο, άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. 18-3 εγκρίνεται. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, τροπολογίες αναφέρει θα τα κατά αποχές εγκρίνονται. Έτσι καταπίπτει 5 η απόφαση για την απαλλαγή. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα αυτής της ψηφοφορίας 19 προς 2 Ευχαριστώ. 6 υπέρ κατά εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά εγκρίνεται, α συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά εγκρίνεται, 14 υπέρ κατά εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά εγκρίνεται, Β συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 21 πέρα στο ελέγχο 14-8 εγκρίνεται C υπέρ κατά εγκρίνεται. D υπέρ κατά εγκρίνεται. D έλεγχος. Πέρας του ελέγχου 17 προς 5 εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ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 G συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται H συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται J υπέρ κατά εγκρίνεται 53 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται J συμβαστική εγκρίνεται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 υπέρ τα αποχές εγκρίνονται το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία αρχιετή ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 17 5 προς 3 Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ Τώρα Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τροπολογία 1 και 4 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 3 κατά καταπίπτει ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την απαλλαγή την ψηφοφορία ονομαστικά πέρας ψηφοφορίας 17 προς 5 το ψήφισμα τώρα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά έλεγχος για την 8 πέρας του ελέγχου εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 σε τρία τμήματα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 όχι. Η 12 καταπίπτει. Συγγνώμη, και η 13 καταπίπτει, λέει πρόεδρος, η 14 επίσης καταπίπτει. Όχι, η 14 δεν καταπίπτει. 14 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 15 υπέρ. Όχι, 15 καταπίπτει, συμβαστική A, υπέρ κατά εγκρίνεται. 18 και 19 και 20 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ αποχές εγκρίνεται β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 με ναι, ψηφοφορία τμήματα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται D συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 31 έλεγχος. Πέρα του ελέγχου εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 38 υπέρ χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας 18 προς 3. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ερχόμαστε στην Επιτροπή των Περιφερειών. 1 και 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Mm αποφασία την απαλλαγή. Όχι, τροπολογίες ένα και δύο έλεγχος. Έλεγχος για την ένα και δύο Πέρας του έλεγχο 16 προς 6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 Πέρα το έλεγχο Απορρίπτεται. 27 σε δύο τμήματα. Περ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Το καταπληκτικό δεύτερο τμήμα. 28 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για την 30. Εγώ πιστεύω ότι έγινε δεκτή, αλλά ας κάνουμε τον έλεγχο. Παρακαλώ. Πέρα στο ελέγχου εγκρίνεται. 31 πίπτη 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πια για τη 37 έλεγχος, έλεγχος της 37. 16 προς 6, 30 38 καταπίπτει, 39 καταπίπτει, 40 καταπίπτει, 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 χωρίς την προφορική τροπολογία ΕΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται 43 ΕΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται 44 ΕΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 16 προς 5 ευχαριστούμε και τώρα θα έρθουμε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβήτη, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. 1, 2, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η απόφαση για την χορήγηση απαλλαγή ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία, 19 προς 3, τροπολογία παριθμών 5, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 6 παρακαλώ 6 Ωραία λοιπόν, εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ,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 όχι, για την 21 πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. πίπτη και το internal 25 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 26 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται το 27 χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύ. Η συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά. Έλεγχος για την 31 παρακαλώ. 31. Έλεγχος, πέρας του ελέγχου εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας, 18 προς 3. Και τώρα θα έρθουμε στο τελευταίο σημείο της ψηφοφορίας. Ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. 1 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η απόφαση για την απαλλαγή ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 19 προς 3, το ψήφισμα ε, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά έλεγχος για την 7 παρακαλώ υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τις τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ Αμπλοκ 2 έως 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Και τώρα θα έρθουμε στη τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστικά άρχια η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες, 18 προς 3, με μία αποχή. Θέλουμε να συγχαρούμε τον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Και τώρα Φτάσαμε στη λήξη τη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πειθαρχία που δείξατε. Την προσεχή Δευτέρα έχουμε την, και πάλι την Επιτροπή. Θα ήθελα να διακόψω εν συντομία τη συνεδρίαση, γιατί θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με τα σημεία υπαριθμών 59, τη μελέτη για τα trust funds. Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf nach einer kurzen Λοιπόν, να συνεχίσουμε τις εργασίες μα. Λοιπόν, έχουμε το σημείο 59 στην μέση διάταξη. Μία μελέτη για τον έλεγχο των καταπιστευμάτων της Ένωσης. Έχουμε το ΣΕΠΣΤΑ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μελετών. Η κυρία Σμιτ είναι η συγκεντριά μας και να δώσω λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Νούνε ή στον κύριο Καρέρα για την παρουσίαση τη μελέτη. Καλώ ήρθατε. Ποιο θα ξεκινήσει, Κύριε Καρέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να μοιραστούμε μαζί σας και να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη που μας ε, εμπιστευθήκατε, που χρηματοδοτεί η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Θεμάτων. Το θέμα είναι πολύ τεχνικό και περίπλοκο και λεπτό. Και ο συνάδελφος ο Χόρχε θα με βοηθήσει. Ο Χόρχε Νούνιεθ Φερέρα. Είμαστε οι ανεξάρτητοι ερευνητέ που κάναμε αυτή την έρευνα. Κάνει μια συγκριτική μελέτη της ε, εποπτείας και των ε, ενωσιακών καταπιστευμάτων και τη διευκόλυνση για τους ε, πρόσφυγες στην Τουρκία. Μας ενδιέφερε η προστιθέμενη αξία για να υπάρχει καλύτερη κανονιστική λειτουργία της Ένωσης. Και ιδιαίτερα ασχοληθήκαμε με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι τμήμα της ε, δημοσιονομικής αρχής για αυτά τα καταπιστεύματα. Και επίσης εξετάσαμε το δικαίωμα της ε, χρηστής διοίκησης που είναι εντός ε, της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η μελέτη αυτή δεν είναι έλεγχος, δεν είναι ποιοτικό έλεγχος συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ασχολείται με την διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την εποπτεία των χρηματοδοτικών δομών, μέσων και μηχανισμών. Λοιπόν, να η μεθοδολογία μας. Κάναμε μελέτη των κειμένων, κάναμε και συνεντεύξεις. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που μας έδωσε τη δυνατότητα να μάθουμε τι προκλήσεις, τι θέματα χειρίζονται και πώς λειτουργούν αυτά τα καταπιστεύματα. Μάθαμε πολλά και από διεθνείς οργανισμούς και μη καπαόμικρον που συμμετέχουν άμεσα στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και είχαμε και μια ομάδα εστίασης, ένα focus group με το οποίο συζητήσαμε και κάναμε ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων. Έχετε ένα πίνακα που παρουσιάζει τα πέντε ταμεία, τα πέντε καταπιστεύματα που μελετήσαμε το καταπίστευμα για την ε, Κολομβία, το Ταμείο για την Αντιμετώπιση της Μετανάστευσης από την Αφρική, την ε, δομή για την Τουρκία που έχει ειδική δομή, το καταπίστευμα Μαντάτ για τη Συρία και το Μπεκού. Το καταπίστευμα Μπεκού. Ένα από τα στοιχεία που εξετάσαμε αναλυτικά είναι πως αυτά τα τόσο διαφορετικά τα πιστεύματα και το καθένα είναι πολύ ιδιαίτερο στην προέλευση, στη φύση, στη δομή. Εξετάσαμε πώς δημιουργήθηκαν πολύ προσεκτικά. Στο άρθρο 187 του Δημοσιονομικού Κανονισμού υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία αυτών των καταπιστευμάτων. Μεταξύ αυτών, η πρώτη ε, προϋπόθεση αφορά μια επίγουσα ή μεταεπίγουσα κατάσταση. Και επίσης πρέπει να υπάρχει θεματική στόχευση και να προσθέτουν αξία σε αυτά που ήδη υπάρχουν στο διεθνέ πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική προϋπόθεση αυτή για το εάν και κατά πόσο είναι σωστό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο καταπίστευμα. Κυρίως βεβαίω έχουν πολύ μεγάλη ευελιξία, είναι το χαρακτηριστικό τους. Αυτό έχει και υπέρ και κατά και τους δίνει και μεγάλη ορατότητα. Δημιουργήθηκαν σε εποχές κρίσης, ιδιαίτερα μετά το 2015, δημιουργήθηκαν μια σειρά από τέτοια καταπιστεύματα για να ανταποκριθούν σε διάφορες κρίσεις. Δίνουν ε, ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτά. Η Επιτροπή παίζει ρόλο κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. Και τα κράτη-μέλη και ένα βασικό πόρισμα αυτή τη μελέτη, επί του οποίου θα αναφερθώ περισσότερο, είναι ο αμεληταίο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Αυτά τα ενωσιακά καταπιστεύματα είναι τα πιο κατάλληλα όργανα για να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Υπάρχει πιστική ανάγκη να δημιουργηθούν και νέα τέτοια. Με βάση τα απορίσματά μας αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να αποτιμηθεί πολύ συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ελεκτικό συνέδριο με το οποίο μιλήσαμε για αυτή τη μελέτη δημοσίευσε μια έκθεση για το καταπίστευμα Μπεκού και ναι μεν κατέληξε ότι λειτουργεί σωστά και είχε έννοια δημιουργία του αλλά πρότεινε στην Επιτροπή να κάνει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση για το εάν και κατά πόσο οι προϋποθέσεις δημιουργίας αυτού του καταπιστεύματος ε, πληρούνται. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για το καταπίστευμα για την Αφρική που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει μια επίγουσα ανάγκη. Και η μελέτη μας θέτει το ερώτημα ποια επίγουσα ανάγκη προέκυψε το 2015 διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει να κάνει με τη μετανάστευση μέσω της Μεσογείου. Μα ήδη υπήρχε αυτή η έκτακτη κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια έναντι της Ιταλίας. Επίση, η, να αντιμετωπίζεται η μετανάστευση ως ε, ένα θέμα έκτακτο, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ε, ανάπτυξης, είναι λάθος ε, υπόθεση. Αυτό έχουμε πολλέ πολλές μελέτε μελέτες που τονίζουν ότι η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων που προκαλούν τη μετανάστευση είναι ένα μακροπρόθεσμο και βασικό θέμα. Δεν είναι κάτι που θα αντιμετωπιστεί με βράχυπρόθεσμες ενέργειε. Τώρα για τη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Εμείς περιγράφουμε πώς ε, δικούνται τα ταμεία αυτά. Το Κοινοβούλιο, όπως είπα, δεν έχει ρόλο παρατηρητή. Καλείται σε συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ε, συναντήσεις των Στρατηγικών Συμβουλίων. καμιά φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λόγω θεμάτων ε, άλλων που είχε να αξιοποιήσει, να αντιμετωπίσει και να ασχοληθεί, δεν χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα τόσο ενεργά όσο θα έπρεπε. Οι λειτουργικές επιτροπές συζητούν τα διάφορα προγράμματα που θα προωθήσουν τα καταπιστεύματα και το θέμα που μας απασχολεί είναι πώς φτάνουν οι προτάσεις σε αυτές τις λειτουργικές επιτροπές. Γιατί υπάρχει κάποια ασάφεια όσον αφορά τα κριτήρια για την επιλογή των ε, εγχειρημάτων. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας. Και αυτό μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους που θα ήθελαν να συμβάλλουν ιδιαίτερα μικρότερες μη καπαόμικρον. Επίσης η μελέτη τονίζει ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ρόλου που παίζουν ως ε, χορηγοί τα κράτη-μέλη και ως ε, ε, φορείς που εφαρμόζουν τα προγράμματα δεν είναι πολύ σαφής. Θέτει το θέμα λοιπόν ενδεχόμενης σύγκρουσης σύμφωντων. Πώς μπορούν να αποφευχθούν, τι μηχανισμούς έχουμε για να τους προλάβουμε. και κατά πόσο είναι κατάλληλα τα καταπιστεύματα αυτά. Αυτοί που εφαρμόζουν καταπιστεύματα είναι οι καλύτεροι, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία προωθούν. Η μελέτη εξετάζει το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας που αναφέρεται σαφώς στις συνθήκες μας και που ε, είναι ένας ρόλος με τον οποίο ε, ασχολείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξετάζουμε διάφορα στοιχεία της δημοκρατικής λογοδοσίας εξάντε, κατά τη διάρκεια και εξ Και δεν θα σας εκπλήξει ότι η μελέτη καταλήγει ότι η εξάντε λογοδοσία είναι χαμηλού επίπεδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υιοθετήσει μη δεσμευτικά ψηφίσματα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ούτε τους στόχους, ούτε το πεδίο εφαρμογή αυτών των ταμείων. Το Κοινοβούλιο βεβαίω ενέκρινε στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό αυτή την δυνατότητα να δημιουργεί καταπιστεύματα. Αλλά μία από τις συστάσει μας είναι ότι με βάση τα πορίσματά μας θα πρέπει να το ξαναδεί το κοινοβούλιο αυτό. Να ξαναδεί και τα αίτια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων δημιουργούνται ούτω ώστε να υπάρχει περισσότερος δημοκρατικός έλεγχο σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ή θα κληθεί ως παρατηρητής ε, διάφορες ε, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μελέτη έγινε το 2017, αλλά δεν έχει επίσημο καθεστώς ε, παρατηρητή με βάση τα καταστατικά αυτών των καταπιστευμάτων. Και αυτό έχει ανησυχήσει και έχει εκφραστεί αυτή η ανησυχία από διάφορε επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Τόνισαν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά τα στρατηγικά συμβούλια. Εκ των υστέρων λογοδοσία. Βεβαίω, ενημερώνει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έρχεται συχνά να παρουσιάσει τα αποτελέσματα διαφόρων προγραμμάτων, κάνει εκθέσεις προόδου και το Κοινοβούλιο λαμβάνει και τους ετήσιους ισολογισμούς και ετήσιες εκθέσεις των καταπιστευμάτων. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να μπούμε στις λεπτομέρειες του κάθε καταπιστεύματος. Σας ενημερώνω ότι η μελέτη δίνει αναλυτική παρουσίαση αυτών που συμμετέχουν στην εφαρμογή των ενεργειών των καταπιστευμάτων. Αναφέρεται στις θεματικές τους προτεραιότητες. Ίσως μετά στο διάλογο μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα και μόνο. Η διευκόλυνση για την Τουρκία, που τυπικά δεν είναι καταπίστευμα. Αλλά παρόλα αυτά, τη μελετήσαμε. γιατί εγκρίθηκε για να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή ε, προσφυγική κρίση. Αν δούμε ποιοι συμμετέχουν στην εφαρμογή των ενεργειών του προγράμματος, θα δούμε ότι οι περισσότεροι είναι εθνικές αρχές και διεθνείς αναπτυξιακές αρχές και ΜΚΟ. Μία από τις κυρίες προκλήσεις είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι εθνικοί φορείς θα χρηματοδοτήσουν με σωστό τρόπο την ε, ανεξάρτητη εργασία των μη κοιόμετρων που να μπορούν να επικρίνουν και τον τρόπο που λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα το ηλεκτρικό συνέδριο δημοσίευσε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την Τουρκία, το κράτο δικαίου, τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και κατέληξε ότι είναι πολύ δύσκολο με τι συνθήκε που ισχύουν να διασφαλίσουμε ότι η διευκόλυνση αυτή ε, επιτυχάνει του στόχου τη και ε, επιτρέπει ε, να επιτευχθούν οι στόχοι της προσπάθειας. Το καταπίστευμα για την Αφρική είναι επίσης ενδιαφέρον. Και αυτό δημιουργήθηκε να αντιμετωπίσει την ε, προσφυγική κρίση. Εστιάζει όλο και περισσότερο στη διαχείριση της μετανάστευσης. Ιδιαίτερα στον διάδρομο της Βόρειας Αφρικής. Και εκεί τίθεται το θέμα της, ε, των προϋποθέσεων που ισχύουν. Δηλαδή το χαρακτηριστικό του είναι ότι βλέπετε τα Υπουργεία Εσωτερικών να υπησέρχονται όλο και περισσότερο στο αναπτυξιακό θεματολόγιο. Δηλαδή θέτουν θέματα αρχών του Υπουργείου Δικαιοσύνη και Εσωτερικών, των Υπουργείων Δικαιοσύνη και Εσωτερικών, τα οποία παρεμβαίνουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τι ρόλο παίζει η Ευρώπη, για παράδειγμα στην Αιθιοπία που είναι από τους κύριους ε, ωφελούμενους. Έχουμε ένα κοινό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και είναι πολύ σαφές ότι συσχετίζεται αυτό με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Απαιτούμε από την Αιθιοπία να λάβει μια σειρά μέτρων ελέγχων, ελέγχου της μετανάστευσης. Λοιπόν, ποιες είναι οι ευρύτερες ε, επιπτώσεις αυτής της ε, διαδικασίας καταδεικνύουμε ότι υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ των καταπιστευμάτων και των ε, πολιτικών προτεραιοτήτων ε, της Ένωσης που ε, είναι ιδιαίτερα επίμαχες και πρέπει να τις εξετάσει το Κοινοβούλιο. Τα καταπιστεύματα σε αυτές τις περιοχές είναι το κεντρικό μέσο ούτω ώστε να παρέμβει στην εξωτερική πολιτική ένωση. Είναι η άσκηση εξωτερική πολιτική μέσω χρηματοδότηση. Χρηματοδοτούν ε, διαδικασίες για την, για διαχείριση της μετανάστευσης εφαρμόζουν ε, και εκτός της Ένωσης τις πολιτικές των Υπουργείων Εσωτερικών. Δεν συμμετέχει όσο θα έπρεπε λοιπόν η Ένωση, όσο θα έπρεπε. Άρα αυτό δεν ε, συνάδει με αυτά που λένε οι συνθήκες για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η εξωτερική και η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Γιατί προχωράμε μόνο με βάση τις έκτακτες και επίγουσες καταστάσεις. Αυτό δημιουργεί προβλήματα για την εφαρμογή των συνθήκων της Ένωσης υπάρχει αυτή η τάση μη δεσμευτικών μέσων τα οποία είναι εκτός συνθήκων και εκτός ενωσιακού προπολογισμού. Εκτός συνθήκων σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν συμμετέχει στη συζήτηση. Για παράδειγμα, στην εταιρική σχέση με την Αφρική. Υπάρχουν μια σειρά από πολιτικά μέσα που έχουμε εγκρίνει με ορισμένες αφρικανικές χώρες για την επανεισδοχή, δηλαδή την απέλαση παρατύπων μεταναστών. Αυτό γίνεται μέσω μέσων που δεν είναι νομικά δεσμευτικά και είναι εκτό συνδικών. Για παράδειγμα, η δήλωση Ένωση Τουρκία. Δεν είναι διεθνή συμφωνία. Και ακόμη είναι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και δεν ξέρουμε ποιο την έκανε αυτή τη δήλωση. Αλλά έχει συνδυαστεί με, αυτό, με αυτή τη διευκόλυνση για του πρόσφυγε. Που είναι πολλά λεφτά για να εφαρμοστεί κάτι που ακόμη συζητάμε περί της φύσης του και επί το οποίο έχει εκφράσει πολλές ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η ιδέα της ανταλλαγής ανάπτυξης μέσω μετανάστευσης. Η μελέτη μας λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Αυτό το στόχο, να αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια για να μειωθεί η μετανάστευση. Οι εργασίες μας λένε ότι είναι λάθος αυτή η σύνδεση. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αποτιμηθούν προσεκτικά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βασικά αίτια που είναι αναπτυξιακά θέματα. Θα πρέπει να αποσυνδεθούν από τον έλεγχο τη μετανάστευση. Είναι μια στρατηγική τη Ένωση. Δίνουμε δισεκατομμύρια σε χώρε όπω η Τουρκία. Ε, τι εντύπωση δίνει έτσι η Ένωση. Είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι στην πολιτική βούληση χωρών όπω η Τουρκία. για να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα που κανονικά θα έπρεπε να είναι ενδοενωσιακό. Δίνουμε λεφτά στην Τουρκία για να κάνει τη δουλειά μα. Αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να ελέγχεται πιο δημοκρατικά. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο μου Χόρχε που θα μας, σας μιλήσει για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να σα πω κάποια συμπεράσματα που έχουμε ξεχάσει από κάποια άλλα καταπιστεύματα. Ε, βέβαια δεν υπάρχει συγκρισιμότητα. Μια που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά, την άλλη μεριά έχουμε άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε καταπιστεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, έχουμε κάποια από ε, τα μέσα διευκόλυνσης για εξωτερική δράση, δηλαδή τα κράτη-μέλη φέρουν κάποια χρήματα, ούτως ώστε οι αναπτυξιακές Τράπεζε και οι ΕΤΕ επενδύουν. Ε, και αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να παρεκτείνουμε αυτή τη χρηματοδότηση, να πετύχουμε κάποια μόχρευση, δηλαδή είναι διαφορετικά καταπιστεύματα. Οπότε παραλληλισμοί δεν υπάρχουν και πολλοί. Έτσι λειτουργούν, μεν, αλλά δεν μπορούσα να βρω κάποια κοινά σημεία εκτός ότι διακρίνονται από μεγαλύτερη διαφάνεια, υποβολή εκθέσεων κλπ. Βέβαια το καθένα έχει άλλο τρόπο λειτουργίας, πολλές φορές ε, έχουν κοινέ εγκαταστάσεις, γραφεία και σχετίζουν τη λειτουργία τους, άρα δεν έχουμε μεγάλη χρησιμότητα. Ε, να ρίξω μια μουσική την Συμπαγκόσμια τρόπο και στον ΟΗΕ και τα σχετικά καταπιστεύματα δεν ναι, διακρίνονται ναι, από υποχρέωση εργοδοσία, έχουν περισσότερου δωρητέ και αντιλαμβάνομεθα δύσκολα και τη λειτουργία του. Έχουμε τώρα και καταστήματα που συγκροτήθηκαν με τη διαδικασία του κατεπήγοντο για συγκεκριμένου λόγου. Μπορούμε όμω να ξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Όπ, είναι άλλη διαφάνεια. Ό,τι δηλαδή Αν δούμε τα διάφορα καταπιστεύματα. Επισημαίνουμε πρόβλημα όποτε έχουμε δωρεά χρημάτων από κάποια χώρα στο καταπίστευμα οπότε η χώρα αυτή μπορεί να επηρεάζει, μπορεί να παρακάμψει τους κανόνες λειτουργίας έχουμε εθνικές πολιτικές που μπαίνουν στο παιχνίδι πάντα σε τέτοιες δωρεές και πάντα ότι υπάρχει προϋπόθεση οι χώρες να διαχειριζονται τα χρήματα και τα θεσμικά όργανα έτσι πετυχαίνουν τους ε, στόχους τους κατά κάποιο τρόπο υφαρπάζοντας το σήμα της φραγίδα ούτως υπήν του καταπιστεύματος Οπότε όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσία, όσον αφορά την εποπτεία, ε, έχουμε σε κάποιε περιπτώσει ε, επίπεδα, αλλά όπως είπαμε συγκροτήθηκαν για συγκεκριμένο έχω και υπάρχουν προβλήματα που χαρακτηρίζουν την πρώτη φάση λειτουργίας. Δηλαδή, υπάρχει μία διαδικτυακή πύλη κοινά γραφεία, οπότε υπάρχει συντονισμός, στενή συνεργασία είναι ευκολότερο ο έλεγχος, ευκολότερο να διαπιστώσει κανείς ποιος τα πάει καλύτερα και ευκολότερη να ζητήσει στοιχείων και πληροφοριών. Άλλως έχουν λοιπόν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια αυτά στοιχεία χαρακτηρίζουν αυτά τα καταπιστεύματα. Μια που συγκεκριμένε απαιτήσει, συγκεκριμένε συνθήκε γέννησαν αυτά τα καταπιστεύματα. Άρα κανεί πρέπει να το εξετάσει και αυτό. Τι γίνεται με το κατέστημα για την Κολονία, για την Κολομβία, συγγνώμη. Και περισσότερα διεθνή καταπιστεύματα έχουν αυτές τις μικτές διευκολύνσεις. Και υπάρχουν μηχανισμοί για τη χάραξη πολιτικής για το μέλλον. Το θέμα είναι όμως για πόσο καιρό θα πηγαίνει έτσι αυτό, γιατί το κατεπήγον δεν διαρκεί πάρα πολύ. Κάποια στιγμή η κατάσταση γίνεται ομαλή, Οπότε γίνεται το θέμα ακριβώ πόσο θα συνεχίσει να υπάρχει το καταπίστευμα. Γι' αυτό και σας λέω, <clears throat> η σύγκριση ήταν δύσκολη. Παρακάτω πάμε τώρα στις τελικές συστάσεις. Πρώτα πρώτα, ο έλεγχος των επιδόσεων της αποτελεσματικότητας ε, της καταλληλότητας σε σχέση με την προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως κανείς να κάτσει και να μελετήσει τι έργο επιτελείται και επίσης ε, όπως είπαμε δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν για πάντα αυτές οι επιδόσεις. Επίσης Έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα το καταπιστήμιο για την Αφρική, αλλά επίσης κάνει και εν μέρει τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Άρα, προσφέρει ο καταπήγον χαρακτήρας του καταπιστεύματος. Κάνει μερικά πράγματα καλύτερα από ότι τα συνήθεια καταπιστεύματα. Εδώ ερωτηματικό. Άρα Όσον αφορά τα καταστατικές συμφωνίες που συγκρότησαν το Ταμείο, θα πρέπει να υπάρχει μία ρήτρα που να αναφέρει τα σχετικά με τους εφαρμοστικούς οργανισμούς, την διακυβέρνηση και τον τρόπο λειτουργίας Οπότε ε, υπάρχουν ερωτηματικά για γιατί να έχουμε κατεξουσιοδότηση συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Για ρίξε μια μαγιά σε παρακαλώ, του συνεργάτη του ομιλητή; Ναι, ναι, ο άλλος κύριος. Ναι, λέμε ότι θα πρέπει αυτούς τους οι καταστατικές συμφωνίες με μεγάλη προσοχή να ορίζουν κάποιο είδους καταρχήν προτίμηση, προτεραιότητα όσον αφορά την κατεξιοδότηση εργασία με τα κρατημέλη, γιατί εδώ υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων με τα κρατημέλη που είτε έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες είτε είναι δωρητές. Ε, ναι, του το δώσω το λόγο γιατί αυτό το διατύπωσε, οπότε και εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν ο κατάλληλος να κάνει την αυθεντική ερμηνεία. Ε, λοιπόν, όπως είπαμε, αυτά είναι τα θέματα της δημοκρατικής υποχρέωσης ε, λογοδοσίας, οπότε υπάρχει το σύστημα του κοινοτικού προϋπολογισμού, άρα όταν τίθεται το ερώτημα του πώς συγκροτήθηκαν αυτά τα καταπιστέματα, ε, βέβαια και είναι σημαντικό να είναι ευέλικτα να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κατεπήγοντα, αλλά πάντοτε κρίνει το ερώτημα του τι γίνεται όταν αλλάξουν οι συνθήκες και τι γίνεται με την δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και επίση για την εξωτερική δράση τα καταπιστεύματα ε, πολλές φορές έχουν κάποιους περιορισμούς ε, χρηματοοικονομικούς μέσω του προϋπολογισμού. Τότε όμως ε, κάνουμε μην παρέξη από τον προϋπολογισμό, οπότε χάνεται η δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας αυτά από οικονομική ανάγκη δεν, δεν περισσεύουν χρήματα ίσως από τον προπολογισμό ή ίσως γιατί χρειάζεται να παρακαμφθεί ο προπολογισμό. Όμως αυτό είναι και το ερώτημα. Λείπουν τα λεφτά. Υπάρχει λόγος να συγκροτηθεί ένα καταπίστευμα το οποίο να λειτουργεί παράλληλα εκτός στο περιθώριο των δημοκρατικών δομών και της λογοδοσίας. Αν να σας συμπληρώσω και εγώ λέω άλλος κύριος αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ακριβώς είναι το θέμα του κόστους διαχείρισης. Υπάρχει η σχετική λεπτομερή μελέτη, δεν είναι πάντοτε σαφής η σχέση ε, κόστους αποτελέσματος της διαχείρισης του καταπιστεύματος. Τελειώσατε, λέει ο κύριος Βόν. Συνεχίζει ο εισηγητής. Αυτέ είναι οι συστάσει μας. Α, για να δούμε. Πούντο, πούντο. Α, να το, να το. Οπότε το επανερχόμαστε στο ότι τι θα γίνει όταν θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες συγκρότησης και Και σε αυτές τις επιχειρησιακές λειτουργικέ επιτροπές το Κοινοβούλιο ανακατεύεται με το δικαίωμα ενημέρωσης και εποπτείας. Και είπαμε θα, η αρχή, το θεμέλιο της μελέτης ήταν η θεσμική ισορροπία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες, να λάβουμε το τι χρειάζεται και έχουμε όλα αυτά τα ε, τα, τα, τα καταπιστεύματα που γεννήθηκαν από το κατεπήγον αλλά πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνθήκη ή οι συνθήκες και αυτό το οποίο πριν συζητήσαμε για το μέσο διευκολύνης με λειτουργία είπαμε ότι πώς είναι δυνατόν να μπορούμε να τα φιλτράρουμε όλα αυτά με τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί το, ο στόχος είναι κάτι το κατεπήγον και επίσης είναι και το θέμα της ανεξαρτησίας των οργανισμών και φορέων που εφαρμόζουν τα σχετικά. Τι γίνεται. Είναι ανεξάρτητες ΜΚΟ, είναι κάποιοι άλλοι φορείς. Έχουν προτεραιότητες διαφορετικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και επανερχόμαστε στις συστάσεις μας και για για τις άλλες, ε, για τα άλλα καταστήματα θα πρέπει να δούμε τι έδρα έχουν, τι γραφεία έχουν και αν υπάρχει κάποια συνάφεια. Και αν το σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτές οι ενιαίες ε, πύλες για τη λειτουργία τους και αυτό δεν μπορούσαμε να το δανειστούμε ως ιδέα και για τα δικά μας καταπιστεύματα στην Ένωση. Και εν κατακλείδη οι συστάσεις μας είναι το ότι θα πρέπει να συνάδουν οι στόχοι με τις γενικές αρχές των συνδικών. Αυτό το διατυπώνουμε και στη μελέτη ότι πολλά από αυτά τα καταπιστεύματα για τα κατεπήγοντα, για το μεταναστευτικό, την Αφρική κλπ. συνδυάζουν ε, εθνικούς πολιτικούς στόχους, ε, τέλος πάντων δικαιοσύνης, ε, δημόσιας τάξης με τους αναπτυσιακούς στόχους. Ακόμα και σε επίπεδο ΟΗΕ έχουν δημιουργηθεί ζητήματα όταν συντρέχουν τέτοιες προϋποθέσεις, τέτοια συμφέροντα για την πολιτική της, ε, την πολιτική τη σχετική χρηματοδότηση. Γιατί εδώ πέρα ανακατεύεται η ανάπτυξη με την ασφάλεια, ε, διαφορετικά πράγματα. Και ξέρουμε από τη θεωρία της διεθνούς αμπισιακής πολιτικής ότι ο συνδυασμός αυτός που είναι προβληματικός. Αλλά θα πρέπει και εμείς να είμαστε συνεπείς με τις ε, αρχές μας, δημοκρατία δηλαδή και ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. όποτε λειτουργούμε σε τρίτες χώρες. Και πάντα να έχουμε κατά νου τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης που τίθενται να αμφισβητήσει. Yeah, yeah, I can. Any more? Is that it? Yes, yes, no, no, that's it, that's it. I that's it. Thank you very much. Sorry, it was the last. Ναι, ήταν η τελευταία σύσταση. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάσετε τη μελέτη σας και το ότι διατυπώσετε τις ε, συστάσεις ε, στο τέλος. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σμιτ. Κύριε, κύριε. Στην κυρία Σμιτ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω τη μελέτη γιατί την έχω διαβάσει. Αν την ε, άκουγα για πρώτη φορά θα ήμουν εντελώ απελπισμένη. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη, δίνει πολλές πληροφορίες, αλλά είναι εξαιρετικ... δημιουργεί και πολλές ανησυχίε. Εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ αυτών των καταπιστευμάτων γιατί αποτελεί έναν γρήγορο και ευέλικτο τρόπο ε, παροχής ε, βοήθειας, ενίσχυσης. Αλλά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι συντάκτες της ε, έκθεσης θέτουν ένα αφιβόλο το μοντέλο του καταπιστεύματος. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια... Δεν θα ήθελα να θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που ανέφεραν ήδη οι συντάκτες της ε, μελέτης, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Ο λόγος για τη δημιουργία των καταπαιδευτευμάτων είναι, όπως σας είπα, μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην ε, κατανομή των κονδυλίων. Αλλά το θέμα είναι από ποιε αξίες εμείς ε, παρετούμεθα όσον αφορά τη διενέργεια δημοκρατικού ελέγχου και την έννοια τη λογοδοσία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, τα, ότι τα καταπιστεύματα μας τα πουλάνε τώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της ταχύτητας ως πλεονεκτήματα αλλά δεν μπορεί κανείς να αποδείξει ότι πράγματι ε, ισχύουν ε, αυτά τα πλεονεκτήματα. Ε, συνέχεια θα πρέπει να θέσουμε ένα σημαντικό ερώτημα. Πόσο σημαντικό είναι στην τομέα της εξωτερικής πολιτικής ε, όσον αφορά τη στρατηγική ε, είναι σημαντικό να προβάλλεται υπό τον όρο ότι παρακάμπτεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm. Επίσης, οι συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίοι αναφέρθηκαν αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, γιατί οι φορείς απόφαση είναι η Επιτροπή και οι χώρες μέλη οι χώρες μέλη ε, προσελκύονται με, με διάφορους τρόπους να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση και αυτό ε, μπορεί να οδηγεί στη στέβλωση όσον αφορά την ε, επιλογή των προγραμμάτων. Και με τον τρόπο αυτό ότι να αμφιβόλω η διαδικασία επιλογής των προγραμμάτων. Ε, κατά πόσο επιλέγουν τα προγράμματα εκείνα τα οποία οδηγούν στη μεριά μιας υπεραξίας. Εδώ πραγματικά υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Και βεβαίως το κόστος της διαχείρισης είναι πολύ ψηλό, άρα για να μιλούμε για μια θετική σχέση κόστος ωφέλειας ε, δεν, ε, δεν συντρέχουν από, από λόγοι. Ε, τώρα, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις και είναι ορατή μια υπεραξία ε, πέρα από τα όρια των ήδη υφιστάμενων εργαλείων. Ε, εδώ θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα κατά πόσο η ανάλυση αυτή δεν ε, κατέληξε μια τυπωμένη διαδικασία από την πλευρά της Επιτροπής. Γιατί περιοριζόμαστε σε άτυπες σημειώσεις και σε συνομιλίες που αντικαθιστούν τελικά μια επίσημη τυπική διαδικασία. Όσον αφορά την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική, ε, πώς θεωρούμε ότι δημιουργείται αυτή η ορατότητα ε, εάν ε, ε, συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες οι οποίες καταλήγουν οι εκθέσεις αυτές, ε, διαπιστώνουμε ότι είναι ελάχιστοι οι πολίτες οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Θεωρώ ότι με την δημιουργία αυτών των καταπιστευμάτων υπονομεύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, το κατά πόσο είναι υπέρ των χωρών ε, μελών και της Επιτροπής. Εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να μην παρακάμπτεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν εξασφαλίζεται ο δημοκρατικός ε, έλεγχος. Ε, και θεωρώ ότι κατά την άποψή μου θα ήταν χρήσιμο οι συνεδράσεις αυτές να γίνονται στο Στρασβούργο ή τις ε, Παρασκευές ή με τους τοπικούς ε, φορείς, ε, για παράδειγμα, στο, στην Πογκοτά, γιατί δεν είναι δύσκολο να αποσταλούν εκεί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Και θα πρέπει βεβαίως οι χώρες μέλη να εκπροσωπούνται στα καταπιστεύματα αυτά όπως έγινε στο Πεκού όπου η Γερμανία και η Γαλλία απέστειλαν τους δικούς τους εκπροσώπους στην Επιχειρησιακή Επιτροπή. Τώρα για το καταπίστευμα της Κολομβίας σύμφωνα με την έκθεση συστάθηκε λόγω παρέμβαση της Ισπανίας. Η ανάγκη δημιουργία ενός τέτοιου καταπιστεύματος για την Συρία προευλήθη εκ μέρου της Επιτροπής. Ερώτημα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μη περαιτέρω δημιουργία άλλων καταπιστευμάτων ε, γιατί απλώς και μόνο επειδή μια χώρα θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό εκπροσωπούνται καλύτερα τα συμφέροντά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, θεωρώ ότι και εδώ υπάρχουν ε, προβλήματα ε, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τις επιχειρησιακές επιτροπές και την λήψη αποφάσεων. Ε, δεν είναι σαφές του πώς προωθούν διάφορα μοντέλα και βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγονται. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτήματα τα οποία μετά την εκπόνηση αυτή της μελέτης παραμένουν πιο ανοιχτά από ποτέ. Ε, και εφόσον πρόκειται κονδύλια των χωρών μελών, τι πρέπει να γίνει, πού βρίσκεται η υπεραξία αυτών των κατατίστευμάτων Και για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα της ευελιξίας, εάν η ευελιξία αυτή δεν ε, λειτουργεί και με άλλα εφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η υπεραξία, γιατί θα πρέπει να δημιουργούνται αυτά τα καταπιστεύματα. Κατά την άποψή μου ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο έχουν νόημα τέτοιου είδου καταπιστεύματα. Η έρευνα δείχνει ότι η Επιτροπή και οι χώρες μέλη θέλουν να δώσουν τα χρήματά τους ταχύτερα και με καλύτερη ευελιξία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ε, ποια κατεπίγουσα ανάγκη υπάρχει εδώ δημιουργίας αυτών των ε, καταπιστευμάτων εφόσον ε, υπονομεύεται ο δημοκρατικός έλεγχος, ε, η άσκηση του δημοκρατικού έλεγχου εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδης ηγητές, αλλά εφόσον αυτοί δεν παρήσανται εδώ, θα ήθελα να κλείσω εδώ με, τις, με την παρατήρησή μου αυτή. Ναι, δεν είμαστε και πολλοί, αλλά ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Να δώσουμε στην Κομισιόν το λόγο για να απαντήσει σε μερικά από τα σημεία που κάνατε. Αλλά πρώτα όμως θα δώσω λόγο στον κύριο Ζέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους συντάκτες αυτής της έκθεσης. Δυστυχώς επιβεβαίωσαν όλες τις επιφυλάξεις που είχα εγώ για αυτά τα καταπιστεύματα. Για μένα αυτοί οι οργανισμοί ήταν ένα μέσο για να ακυρωθεί η δυνατότητα ελέγχου μέσω του Κοινοβουλίου, όπως γίνεται και με το Αναπτυξιακό Ταμείο. Και όλα όσα μας υποσχέθηκαν και κάποιοι συνάδελφοι τους πίστεψαν. Τελικά δεν ισχύει. Για παράδειγμα, το, ταμείο, το καταπίστευμα για την Αφρική. Ήταν απόφαση των κρατών μελών στην Λαβαλέτα. Λόγω της, ε, του προσφυγικού. Θέλαν να γίνει κάτι στα γρήγορα. Για να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική πίεση που δεν ξεκίνησε το 2015. μετά το τραγικό ατύχημα της Λαμπεντούζα που είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ε, δημοσιότητα. Ήθελαν να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Αλλά τι κατεπίγουσα, τι έκτακτη ανάγκη. Δεν υπήρχε καμία έκτακτη ανάγκη. Δημιουργήθηκε το 16 για να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση. Το 90% της χρηματοδότησης είναι από το Αναπτυξιακό Ταμείο, το EDF και από τμήματα του προπολογισμού, του γενικού προπολογισμού και κατά 10% είναι συμβολές κρατών μελών της Νορβηγίας και της ε, Ελβετίας. Και από ό,τι έμαθα, οι χώρες αυτές θέλουν μέσω της συμβολής τους να χρηματοδοτηθούν ε, προγράμματα τα οποία ήδη είχαν σχετιστεί με αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Το EDF και γενικά οι πόροι για την αναπτυξιακή πολιτική στο γενικό προπολογισμό μας υπόθηκε πάντα ότι θα χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα, μακρόπνοα προγράμματα για να υπάρξει ανάπτυξη σε κάποιες χώρες του κόσμου που χρειάζονται φυσικά ανάπτυξη. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι μπορούμε από αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους παίρνουν δισεκατομμύρια. Τίθεται λοιπόν ήδη το ερώτημα, ήταν λάθος προγράμματα, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν, δεν μπορέσαμε να το οδηγήσουμε εκεί που θέλαμε. Τα παίρνουμε, τα δίνουμε σε αυτά τα καταπιστεύματα για να αντιμετωπιστεί απευθεία η μεταναστευτική κρίση. Και μετά από δύο χρόνια λειτουργίας αυτού του καταπιστεύματο είναι ακόμη στη φάση υπογραφής ε, συμβολέων και 50% περίπου των πόρων που δόθηκαν σε αυτό το καταπίστευμα επιστρέφουν στα κράτη-μέλη ή σε διάφορου αναπτυξιακού οργανισμούς ή σε άλλους διεθνεί οργανισμούς που δεν ξέρουμε τι κάνουν και δεν τους ελέγχουμε. Όλα αυτά για μένα είναι απολύτω παράλογα. Και καταλαβαίνω και εκπροσώπους ε, οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών που υποτίθεται ότι βοηθάμε που με ρωτάνε. Είχατε μια συνάντηση κορυφή το 2015 όπου όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν να μα βοηθήσουν γιατί δεν βλέπουμε τίποτα από όλα αυτά μετά από δύο-τρία χρόνια επιτόπου. Και έχουμε διάφορες ε, οργανώσεις που με αυτόν τον τρόπο διευρύνουν την δραστηριότητά τους. Στην ουσία λοιπόν είναι ένας αυτοτροφοδοτούμενος μηχανισμός γραφειοκρατικός ε, που λειτουργεί με βάση ό,τι κάναμε πριν, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Οι χώρε όμω αναπτυσσόμενε θέλουν εντελώ διαφορετική αναπτυξιακή κατεύθυνση από αυτή που του δίνουμε. Δεν βρίσκω λόγια για να τα εκφράσω όλα αυτά. Και η μελέτη αυτή ακριβώς επιβεβαιώνει αυτή την άποψή μου. Πρέπει να γίνει μια θεμελιώδης ε, αλλαγή κατεύθυνσης. Να διατυπώσουμε στόχους οι οποίοι να μην βαλτώνουν ε, μέσα στη γραφειοκρατία Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αναπτυξιακή πολιτική. Να βοηθάει επιτόπου εκεί τον πληθυσμό και να υπάρχει και ενίσχυση των ε, δημοκρατικών δικαιωμάτων ε, και όχι απλώς να θεριεύουμε τη γραφειοκρατία η οποία λειτουργεί ως αυτός σκοπός. Ελπίζω η μελέτη να συμβάλλει να προχωρήσει αυτή η συζήτηση και να δούμε την κατεύθυνση της ε, αναπτυξιακής μας πολιτικής. Για παράδειγμα το EDF προβλεπόταν για τα κράτη που είχαν ε, συμμετάσχει στην Συμφωνία Κοτονού Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ Τώρα όλα αυτά γίνονται μέσω του καταπιστεύματος, όπου συμμετέχουν και τα κράτη της Βόρειας Αφρικής ή άλλα κράτη. Οπότε τίθεται το ερώτημα, μα πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Νομίζω ότι έχουμε επαρκή τεκμηρίωση, ούτως ώστε να να διεξαγάγουμε αυτή τη συζήτηση μέσω αυτής της μελέτης. Αλλά πρέπει να την κάνουμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Okay, Ευχαριστώ κύριε Ζέλε. Λοιπόν, νομίζω τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρεις θέλουν το λόγο. Η κυρία Φερνάνα από την Γενική Δευσυνία, η κυρία Μοντέζη από την ΤΕΦΚΟ και ένας συνάδελφος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Μπριγκόντι. Η κυρία Φεράν πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι, θα ξεκινήσω εγώ. Μοντέζη από την ΤΕΦΚΟ. Ευχαριστούμε κύριε Βουλευτέ και εσά κύριε Πρόεδρε και εσεί κύριε Σύμβουλοι για την ανταλλαγή απόψεων. Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο σε σχέση με το εύρος αυτών των ε, θεμάτων που συζητούμε οπότε ακριβώς όπως είπε και ο εισηγητής προσβλέπουμε σε άλλες ευκαιρίες για να τα συζητήσουμε και να μπορούμε να εξετάσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας για να μην φύγουμε από εδώ ε, απογοητευμένοι μια που δεν δόθηκε αρκετός χρόνος για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν και ευχαριστούμε τους συμβούλους και πάλι για την μελέτη και θα πρέπει να πω ότι θα προτιμούσαμε εμείς έναν οικονομικό έλεγχο για τους οικονομικούς ελέγχους μπορούμε να αντιδράσουμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένες διαπιστώσεις. Όμως δεν ισχύει εν προκειμένου αυτό. Τα είπαμε στην προπαρασκευαστική φάση, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τα συμπεράσματα, ούτε να εισφέρουμε κάποιο είδους ε, στοιχεία τα οποία θα διόρθωναν κάποια σημεία. Πάντως, αν θέλει το Κοινοβούλιο, εμείς ευχαρίστως να απαντήσουμε όσον αφορά κάποια λάθη, κάποιες ανακρίβειες της μελέτης. Για να δούμε τώρα κάποια σημαντικά σημεία που αναφέρθηκαν. Ελπίζω θα υπάρχει ευκαιρία να επανέλθουμε σύμφωνα με ό,τι αποφασίσει το Κοινοβούλιο ως συνέχεια της προβληματικής που θα ξεκινήσει. Ε, βέβαια δεν μπόρεσε η μελέτη να λάβει υπόψη ούτε κάποια δεδομένα τα οποία αφορούν τις ε, εκτελεστικές εκθέσεις του 17 γιατί είχαμε εκεί σημαντικά βήματα πρόοδο άλλωστε αυτά τα στοιχεία είναι δημοσιοποιημένα στο ίντερνετ στα σχετικά Οπότε, γενικώ υπήν να ευχαριστήσουμε τους συμβούλους οι οποίοι τελικά ε, κατέληξαν στο ότι αυτά τα ε, καταπιστέματα είναι σημαντικά μέσα για να καλύψουν τους στόχους μας για δυο βιώσιμη ανάπτυξη και να δημορφωθεί μια γενικότερη συνένεση για αυτούς τους στόχους που συμμεριζόμαστε και συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο. Ε, βέβαια, όπως ελέγχθη, αποδεικνύει από τη μελέτη ότι υπάρχει μια ε, πολυμορφία κατά Πολυμορφία που είναι κάτι το φυσιολογικό, γιατί όπως προβλέπεται από το άρθρο 187 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, προβλέπεται, λέγω, η συγκρότηση πολλών διαφορετικών καταπιστευμάτων. Και έκαστο εξ αυτών καλύπτει κάποιες ανάγκες, αντιστοιχεί σε κάποιους συγκεκριμένους στόχους που έχουν εγκριθεί και προβλέπονται από τα καταστατικά τους και φυσικά το Κοινοβούλιο έχει ελεγκτική αρμοδιότητα επ' αυτών. Το θέμα είναι κατά πόσον όλα τα καταστήματα καλύπτουν αυτά, αυτούς τους στόχους, αν μας δίνουν κάποια προσταμινή αξία, γιατί είπαμε ότι είναι δύσκολο αυτό να αποδεχθεί για όλα τα καταστήματα όπως είπαν και οι για την πρώτη και κάποια καταστήματα που έχουν ε, βέβαια από προβολή πολιτική και θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε εδώ επικαλύψεις με άλλου είδους ε, θεσμικά όργανα. Οπότε είπαμε ότι κάθε καταπίστευμα αντιστοιχεί σε κάποιους στόχους, σε κάποιες πολιτικές και να απαντήσω για το σύνολο των παρατηρήσεων σε σχέση με τις συστάσεις των συμβούλων γιατί η πρώτη σύσταση είχε να κάνει με το πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε το Better Regulation Framework ούτω ώστε έτσι να συγκροτούμε καταπιστεύματα. Και όταν μιλάμε για τέτοιου είδους κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο, ε, μιλάμε για νομοθετικές πράξεις. Και έχουμε πει ότι αυτά τα καταπιστεύματα θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους. Και η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ότι όλα θα γίνουν με κάποιους χρηστή διαχείριση, με διαφάνεια, με αναλογικότητα, με αποτελεσματικότητα, με αποφυγή διακρίσεων. Ε, για όλα αυτά εμείς έχουμε στρατευτεί, έχουμε δεσμευτεί, για όλα τα καταπιστεύματα. Βέβαια δεν μπορούμε τώρα να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες του κάθε καταπιστεύματος, αλλά προσπαθούμε να τηρούνται όλες αυτές οι αρχές της χρηστής διαχείριση. Τώρα όσον αφορά τη συγκρότηση του κάθε καταπιστεύματος επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο γεννήθηκε από την Επιτροπολογία. Και σήμερα με την Επιτροπολογία έχει ελεγκτικό δικαίωμα και αρμοδιότητα το Κοινοβούλιο. Κάποιες δε συστάσεις, για να δούμε την υπαριθμόν 5 ή την υπαριθμόν και αναφέρονται σε αυτόν τον ελεγκτικό ρόλο του Κοινοβουλίου. Και να σας τονίσουμε ότι εμείς προβληματιστήκαμε όταν καταρτίστηκε, όταν συγκροτήθηκε το κάθε ε, διαπίστευμα από εδώ και εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οτιδήποτε θέλει να θέσει το Κοινοβούλιο σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή, ούτω ώστε να παρουσιαστεί η δουλειά η οποία γίνεται σε κάθε καταπίστευμα. Είχαμε την ευκαιρία επανειλημμένα να έρθουμε και να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα, της επιδόσεις, τους στόχους. Οι εκθέσεις που προετοιμάζουμε για τα καταστήματα είναι πολύ περισσότερες από όσες κάνουμε ας πούμε για το ε, Ταμείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. Οπότε γι' αυτό σας λέω τώρα, ήδη ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός έχει τροποποιήσει τι αρμοδίε του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτά που λένε οι συστάσει. Ε, γι' αυτό και ε, είναι ευξημένε οι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου για αυτά τα για, για, για τη συγκρότηση, χρειάζεται η έγκρισή του όσον αφορά τα ε, ταμεία, χρειάζεται μια προηγουμένη διαβούλευση. Πάντως τονίζουμε ότι τώρα υπάρχει αυτή η βούληση της Επιτροπής το Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει και να επιλαμβάνεται για να, να, να πληροφορείται ενδελεχώς για τα των καταπιστεύματων Και υπάρχει αυτό ο ρόλο του παρατηρητού στα διοικητικά συμβούλια. Ε, αυτό βέβαια και πολλέ φορέ είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί. Τα είπε και η κυρία η συγγήτρια. Πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα τόπου, χρόνου, τέλο πάντων. Ε, εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να μην γίνονται διοικητικά συμβούλια την Παρασκευή που είναι δύσκολη μέρα για το κοινοβούλιο. Οπότε, όποτε θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει το Συμβούλιο στην Αφρική, Οπότε αυτό μας φέρνει πιο κοντά στους εταίρους μας. Επίσης προσπαθούμε να εξασφαλιστεί συμμετοχή το Κοινοβουλίου με κάποιο είδους τηλεσυνεδρίαση και να πως υλοποιείται ο ρόλος του παρατηρητή για το Κοινοβούλιο. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επικοινωνία. για κάθε διαπίστευμα, οπότε και έχουμε την ετησία έκθεση που συντάσσεται για κάθε κάτω για το τι έχει γίνει, τι επιδόσεις έχουν σημειωθεί, για τα των λογαριασμών του καταπιστεύματος και εμείς ε, είπαμε με χαρά μας να εμφανιζόμεθα ενώπιον των κοινωνικών επιτροπών για να συζητούμε. Να, είπαμε και για το καταπιστήμα για την ε, Αφρική που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο. Επίση και για τα χρηματοοικονομικά υπάρχει μια εξαμηνία έκθεση την οποία διαβάζουμε στο Κοινοβούλιο. Επομένως, είναι σημαντικές ελεγκτικές αμμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Πάντως, έχουμε τα καταπιστεύματα που είτε γίνονται από τους δωρητές, είτε από κάποιο είδου ε, χρηματοοικονομικά μέσα πολιτική τα οποία δεχίζεται η Κομισιόν. Οπότε με την ευκαιρία να σας ξανατονίσουν ότι άπαξ και αυτά τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα πηγαίνουν στα καταπιστεύματα, τότε υποχρεώνεται η Κομισιόν να δει κατά πόσον όλα αυτά εξυπηρετούν τους σκοπούς του κάθε κονδυλίου, του κάθε οικονομικού εργαλείου, μέσου τέλος πάντων. Ο, οπότε είμαστε πρόθυμοι να προβούμε και να συμμετάσχουμε, να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο για μια ακόμη πιο εντελεχή ανάλυση. Και έτσι θα υλοποιηθεί αυτός ο υποπτικός ρόλος του Κοινοβουλίου. να προσθέσουμε τώρα κάτι όσον αφορά τη σύσταση παριθμών 2 που αφορά τα του καταστήματος της Αφρικής. Γιατί είναι θεματικό καταπίστευμα και συγκροτήθηκε στη βάση του κατεπήγοντος οπότε παραλαμβάνουμε ότι όταν συγκροτήθηκε αυτό το καταπίστευμα να μην ξεχνούμε ότι σοβούσε η κρίση στο Σαχέλ υπήρχε αστάθεια αλλά και στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Είχαμε και την κρίση με την Μπόκο Χαράμ και φυσικά το κοινοβούλιο είχε ιδιαίτερη ευαισθησία για όλα αυτά. Διασυνοριακή κρίση, τρομοκρατικές επιθέσεις στη, στο βόρειο Σαχέλ και πριν το μεταναστευτικό είχαν προταθεί κάποια καταπιστεύματα ούτως ώστε να καλυφθεί το πρόβλημα ασφάλειας στο Σαχέλ και στην περιοχή της λίμνης ε, Τσάδ, γιατί εκεί ακριβώς δρούσε η Μπόκο Χαραμ. Και με το καταπίστευμα. Φτάσαμε στις μέρες του μεταναστευτικού οπότε και λύσαμε και αποφασίσαμε τον Μάρτιο στην ε, Βαλέτα να υπάρξει ε, να συγκριθεί ένα ταμείο για το μεταναστευτικό που υπήρχε στο καταπίστευμα που σας είπα όπως είπαμε έχει πολλούς στόχους το ταμείο για την ε, Αφρική ασφάλεια, σταθερότητα σε Σαχέλ και Λίμνη Τσάδ. Αλλά στόχος είναι και το να κάνουμε κάτι για τις απότερες αιτίες της μετανάστευσης. Να βοηθήσουμε τους ε, μετανάστες κατά τη μετακίνησή τους τελικά να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να εξασφαλίσουμε την επιστροφή όλων αυτών που είναι εκτοπισμένοι, που είναι πρόσφυγες στη σχετική περιοχή. Άρα εδώ υπάρχει μια πανσπερμία ταμείων. Είναι πλούσιο αυτό το θεματολόγιο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την επίγουσα, την πιεστική κατάσταση στο Σαχέλ και στη Λίμνη Τσάδα. Με την ευκαιρία Επίσης, να δούμε και κάτι άλλο. Αναφέρθηκε από τους συγητές, αναφέρθηκε από τους συμβούλους όσον αφορά αυτή την, την ανάμιξη των πολιτικών. Ο κύριος Βον, μήπως θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε σε δύο λεπτά, γιατί ε, εκτός από εσάς και άλλοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι βεβαίως συμπαθάτε με που μακρηγόρησα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ναι, ναι ακριβώ γι' αυτό να δώσουμε και σε άλλου ευκαιρία. Migration. Άρα υπάρχει αυτή η σχέση του καταπιστεύματο με, με τη μετανάστευση με τα άλλα θέματα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είπαμε ότι να μην υπάρχουν επαναπροωθήσει και έτσι μπορέσαμε να σώσουμε σύμφωνα με στοιχεία του 17 σχεδόν 4.000 ε, από κάποιους που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί στην έρημο. Και πάνω από 10.000 γύρισαν στη χώρα τους, οι οποίοι ήταν σε ε, κατάσταση ανάγκη στην ε, Λιβύη. Οπότε να, που καλύπτουμε και το θέμα της μετανάστευσης, αλλά υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την επαναπροώθηση των μεταναστών. Και όλα κάτι θα πρέπει να γίνει για αυτές τις ε, μεταναστευτικές ροές και να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε όσον αφορά το δουλεμπόριο των ε, προσφύγων και την λαθροδιακίνηση. Α, και κάτι άλλο πρέπει να σας πω, το οποίο αναφέρθηκε στη συζήτηση, δηλαδή έχουμε την σύσταση 4 και τη σύσταση 6 όσον αφορά το ρόλο των εκτελεστικών υπηρεσιών των κρατών ε, μελών και των ΜΚΟ είναι σημαντικό. Είπαμε στο καταστατικό των καταπιστευμάτων αναφέρεται το ότι μπορούν να επιστρατευτούν αυτές οι υπηρεσίες των κρατών μελών. Και γιατί, γιατί οι εκτελεστικοί οργανισμοί, για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό που θα αποτελέσει προσθέμενη αξία. να υπάρχει πιο συγκεκριμένη συνεργασία, πιο πολλή αξιοποίηση των γνώσεων, της εμπειρίας των εκτελεστικών υπηρεσιών της κάθε χώρας και έτσι αυτές τις γνώσεις, αυτή την εμπειρία να την αξιοποιήσουμε λέγω ούτω ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε πιο αποτελεσματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι εκτελεστικοί οργανισμοί έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί ρίχνετε μια ματιά τι γίνεται για το Ταμείο της Αφρικής. Υπάρχει εκεί κάποια κατανομή ισομερής. 22% που αφορά τους, ε, τις ΜΚΟ και ένα μεγάλο ποσοστό ταμείων και πόρων που διακινούνται και που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ σε συνεργασία με τη ΜΚΟ. Τώρα υπάρχει το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Τα κράτη, μέλη, καμιά φορά έχουν σχέση με αυτό το φαινόμενο, υποστηρίζουν κάποια προγράμματα ως παρατηρητές. Δεν έχουν ψήφο τα κράτη-μέλη όσον αφορά την λήψη αποφάσεων για αυτά τα καταπιστεύματα. Και τώρα να δώσουμε την σκητάλη στους συναδέλφους. Να σας πούνε για όλα τα μια τελευταία σύσταση. Είναι υπαριθμόν εννέα και αφορούσε αυτά τα, τα, τα κοινά γραφεία. Είναι πολύ σημαντικό να επιστοδεύουμε περισσότερα ταμεία και αυτά να περνάνε από κάποιο είδου κοινή διαχείριση με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα πολιτικής. Γιατί έτσι έχουμε συνοχή, έχουμε συμπληρωματικότητα, έχουμε συνέργεια με τα υπόλοιπα εργαλεία μας, τα υπόλοιπα μέσα πολιτικής. Γιατί δεν έχουμε επικάλυψη. Βέβαια μπορούμε να έχουμε κάποιο είδους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Διακόπτει ο κύριος Βον. Καλά, καλά, καλά. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ. Ε, πολλά υπόθηκαν και πραγματικά προσυπογράφω τα όσα είπε η συνάδελφός μας ιδιαίτερα όσον αφορά την προσθέμενη εξία αυτού, αυτών των καταπιστευμάτων, κάτι το οποίο δεν αναφέρει παρκώς ε, η μελέτη. Τώρα, όσον αφορά τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στη Τουρκία, όπως αναφέρει ορθώς ε, η έρευνα, δεν πρόκειται για ένα καταπίστευμα παρόλο που η γλώσσα ε, σε ορισμένα σημεία της έκθεσης μας παραπλανεί. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, διορθώνουν αυτά τα σφάλματα στην ε, μελέτη. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τα όσα αναφέρθηκαν ε, σήμερα για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Καταρχήν τη διασύνδεση μεταξύ αυτού του εργαλείου και της πολιτικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρησιμοποιήθηκαν, ελέγχθη, συγγνώμη, εδώ το πρωί ότι αυτή είναι μια επιπλέον συνθήκη, μια κάπως έντονη ε, διατύπωση. Ε, θεωρώ όμως ότι η διευκόλυνση ε, αυτή για τους πρόσφυγες δημιουργήθηκε το 2015 και βασίζεται στα 2010 και 2014 της συνθήκης που αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών μελών ε, προκειμένου να υπάρχει αναπτυξιακή συνεργασία ε, συνεργασία στα θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής και της ε, χορήγησης βοήθειας. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια πλατφόρμα συντονισμού εδώ και όπου όλες αυτές οι αποφάσεις εφαρμογής ελαμβάνονται βάσει των τυπικών διαδικασιών επιτροπολογίας σύμφωνα με τα βασικά εφαρμοστικά εργαλεία ε, δηλαδή της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εργαλείου για την πρωταξιακή βοήθεια και θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη ότι δεν μπορούμε να προβούμε στην ε, παραδοχή ότι με τα καταπιστεύματα αυτά υπονομεύεται η διαδικασία της υποτροπολογίας ε, υπό την έννοια ότι η εφαρμογή, η εκτέλεση μάλλον γίνεται σύμφωνα με τις εφιστάμενες ε, διαδικασίες για όλα τα όργανα εφαρμογής. Και ε, όσον αφορά τα δύο δισεκατομμύρια από τις χώρες ε, μέλη, το ποσό αυτό υποβάλλεται στον, στις κανονικές διαδικασίες για τον έλεγχο του προπολογισμού. Άρα υπάρχει μια εποπτεία συνολική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το εργαλείο αυτής της διευκόλυνσης. Εμείς έχουμε προσκληθεί ως παρατηρητές στο Steering Committee και θα προσέξουμε να διενεργηθούν σε ένα χρόνο που θα μπορεί να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εισφορέ των χωρών μελών εντάσσονται στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ε, τα τρία δι υποβάλλονται στην ε, συνήθεια διαδικασία ελέγχου και ε, η Επιτροπή εκπονεί μηνιαία αναφορές Τώρα όσον αφορά το, χώρο, το ρόλο των ε, υπηρεσιών των χωρών μελών και προσυπογράφω πλήρως ε, την παρτίδα τη κυρία Μοντέζη όσον αφορά το ενδιαφέρον το οποίο έχουμε ε, προκειμένου να συνεργαστούμε με τι υπηρεσίε των χωρών μελών όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και επίσης το ίδιο ισχύει και για την συνεργασία με τις ΜΚΙΟ. Υπάρχουν περιπτώσεις βεβαίως ε, όπου οι μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις ε, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φορείς εκτέλεσης. Για παράδειγμα, όταν υποβάλλουν προτάσεις για την δημιουργία ενός νοσοκομείου στην Τουρκία. Όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία οδηγούν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε αφορά την επιλογή αυτών των υπηρεσιών και δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά επιλέγονται ε, σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, ιδιαίτερα εφόσον ενισχύονται, ε, ε, συνδέονται μάλλον με, τα, με την πρωταξιακή διαδικασία, ε, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν ορισμένες υπηρεσίες των ε, χωρών ε, μελών. Αυτές είναι οι βασικές ε, παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Εκτιμούμε πάρα πολύ την έκθεση. Λυπόμεθα που δεν είμαστε σε θέση να δούμε ένα σχέδιο έκθεση ώστε να εκφράσουμε τα δικά μας σχόλια με πιο ακριβή τρόπο ε, κάτι που κάναμε σήμερα αλλά βεβαίως θα είμαστε ευτυχείς να επανέλθουμε στο θέμα αυτό ε, θα πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση στις 12.30 αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους να παρέμβουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να πω ότι παρόλο που η μελέτη δεν είναι μια αξιολόγηση ούτε ένας έλεγχος. Παρόλα αυτά ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, συνολική πραγματικότητα του ε, ποια είναι τα επιτεύγματα των καταπιστευμάτων αυτών μέχρι στιγμής. Αλλιώς αποκρινθούμε από την ουσία του ερωτήματος του κατά πόσο τα εργαλεία αυτά έχουν εκπληρώσει ορισμένου στόχους. Θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι σε σύγκριση με τρία-τέσσερα χρόνια πριν αυτή τη στιγμή ε, ε, υπάρχει καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από ό,τι τρία χρόνια πριν. Υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και υποστήριξη από τις χώρες ε, μέλη όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία στην Κολομβία. Άρα λοιπόν η συνολική αυτή πραγματικότητα θα πρέπει να είναι κομμάτι της ε, αξιολόγησης. Και με αυτό οδηγούμε σε ένα άλλο σχόλιο το οποίο δεν έφερε αφορά το ρόλο των χωρών μελών. εάν είμαστε σε θέση να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα με όρους της καλύτερης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια συντονισμένη, ενοποιημένη δράση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών μελών σε διάφορες ε, πολιτικές ε, πλατφόρμες, ε, την πολιτική ανάπτυξη, την πολιτική εμπορίου και ε, τις ε, πολιτικές που μπορούν ε, να συντονίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες μέλη σε σχέση με τους εταίρους τους. Άρα λοιπόν ε, δεν ε, υπάρχει μόνο η χρηματοοικονομική ε, πτυχή όσον αφορά αυτά τα καταπιστεύματα ή δεν υπάρχει μόνο το στοιχείο της παροχής πραγματογνωμοσύνης αλλά πρόκειται για μια συνολική μόχλευση μια συντονισμένη δράση μεταξύ ενωσιακού επίπεδου και χωρών μελών το οποίο δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε. Επίσης χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση, μελέτη αναφέρεται στο μέλλον προκειμένου να βρεθούν περισσότερες δυνατότητες εντός του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει μια ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή συστασία όσον αφορά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης όπου θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία και μέτρα τα οποία επιτρέπουν εντός του κανονικού προϋπολογισμού να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο συγητής μας ε, ε, συντάκτης έκθεσης πρέπει να πάνε σε μια άλλη συνεδρία, όμως ίσως θα έπρεπε να τους δώσουμε δύο-τρία λεπτά για να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ για όλα σας τα σχόλια και τις ε, φορέ σας, τις αντιδράσεις σας εκτιμούν πάρα πολύ και ε, βεβαίως θα τις λάβουμε υπόψη μας. Ε, το, η εμβέλεια της έκθεσης ήταν η διαχείριση, η διακυβέρνηση και όχι μια ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων, γιατί αυτό προβλέπεται μια νέα μελέτη. Εμεί κάναμε μία ε, ε, ουδέτερη εξολόγηση των θεμάτων της ε, διαχείρισης των, σε σχέση με τα καταπιστεύματα. Βεβαίως, εμείς λαμβάνουμε υπόψη σαν ισχύ, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε την επιστημονική μας ουδετερότητα στο πεδίο αυτό θα δούμε, θα λάβουμε υπόψη τι ε, διορθώσεις και στο μέτρο που δεν στρεβλώνουν τα δικά μας αποτελέσματα θα τις συμπεριλάβουμε. Όσον αφορά την καλύτερη ρύθμιση, αυτό είναι το πρίσμα το οποίο ε, εξετάσαμε με πολύ προσοχή γιατί δεν ασχολούμαστε με νομικά ζητήματα. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Όμπουτσμαν είπε ότι το θέμα της χρηστής διαχείρισης αφορά όλα τα όργανα συμπεριλαμβάνομενης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δήλωση της Επιτροπής ε, δηλώνει ότι ανεξάρτητα από την ε, ε, σχέση αυτή μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίζει ένα νομικό πλαίσιο που να καλύπτει τα τεκτενόμενα. Και αυτή τη στιγμή, εν ώψη των γεγονότων, δεν θεωρούμε ότι αυτό έχει γίνει. Επίσης, όσον αφορά το κράτος ε, δικαίου, και εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή διακυβεύεται το κράτος ε, δικαίου στην ε, Τουρκία και είναι όμοιρος της κυβέρνησης. Όσον αφορά την Αφρική, κάναμε μία case study για την Αφρική και εδώ εξετάσαμε ένα project ε, SIMS που αφορά την ε, παράνομη μετανάστευση και το οποίο διασυνδέει τις αιτίε μετανάστευση με την παράνομη μετανάστευση. Βέβαια, εκτιμούμε το σχόλιο της Επιτροπής ότι υπάρχει μια ανάγκη καλύτερης ε, παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων. Αυτό το οποίο διαλευκαίνει η ε, μελέτη είναι οι προκλήσεις όσον αφορά την δημοκρατική ε, λογοδοσία Βεβαίω η Επιτροπή και το ρόλο του Κοινοβουλίου βεβαίω θα πρέπει να έχει αυτονομία η Επιτροπή, αλλά υπάρχει μεγάλο περιθώριο όσον αφορά τις βελτιώσεις για την συνεχή ε, λογοθεσία σε σχέση με τις ε, αποφάσεις που έχουν ληφθεί και την διαδικασία της επιτροπολογία. Όσον αφορά την διευκόλυνση για την Τουρκία, η μελέτη λέει ότι ε, δεν μπορεί να συγκριθεί με τα άλλα καταπιστεύματα. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Και πραγματικά δεν είναι συγκρίσιμο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο λέει η μελέτη είναι ότι αυτό το καταπίστευμα έχει συνδεθεί με ένα πολιτικό εργαλείο ε, και που ε, δεν έχει γίνει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι το οποίο έχει βαθύτατες επιπτώσεις όχι μόνο για τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία αλλά και τα δικαιώματα των ανθρώπων τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το οποίο λέμε εν συντομία στην ε, μελέτη. Νομίζω αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. ίσως ε, θα πρέπει να συντονίσετε τις προσπάθειές σας και να καλύψετε τα τυχόν ε, λίματα της έκθεσης. Ευχαριστούμε όλους. Ολοκληρώνει τη συνεδρία.